Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε μια ψηφοφορία που θα κρατήσει αρκετά, πιστεύω. Είναι χοντρό το πακέτο, αλλά πιστεύω ότι θα τις ολοκληρώσουμε σύντομα. Λοιπόν, σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξη δεν βλέπω να υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, άρα θεωρώ ότι εγκρίνεται. Έτσι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, ωραία, εγκρίνεται. Λοιπόν, σημείο δεύτερο, έγκριση των πρακτικών. Τα σχέδια των συνεδριάσεών μας για τις 19 Νοεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου και 22 Ιανουαρίου είναι στα εγγραφά σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις ε, για τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών. Όχι. Ωραία. Προτείνω, ως συνήθως, ε, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά εάν δεν υποβληθούν ε, τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Σήμερα έχουμε διερμηνία στις εξής γλώσσες γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά. Ο Συνήθω σας υπενθυμίζω ότι η συνεδρίαση είναι στο διαδίκτυο. Αποφάσεις των συντονιστών της 4 Φεβρουαρίου 2019. Οι αποφάσεις των συντονιστών της 4 Φεβρουαρίου 2019 σας ε, απεστάλησαν στις 5 Φεβρουαρίου με mail και θα θεωρηθεί ότι ανακρίθησαν επισήμω εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της 8 Συγγνώμη, εφόσον ε, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου δεν υποβλήθησαν αντιρρήσει και γι' αυτό ε, θεωρείται ότι ανακρίθησαν. Έχουμε 13 ε, εκπρόσωποι από την Ομοσπονδιακή Οργάνωση Νεολαίας οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την ψηφοφορία για το έρασμο ΣΥΝ. Σας ε, καλωσορίζω και ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα η παραμονή σας στις Βρυξέλλε. Τώρα, να σας ενημερώσω ότι επειδή δεν υπευλήθησαν ε, αντιρρήσει για το σχέδιο έκθεσής μας για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα μέτρα επίγουσης ε, καταστάσεω για το έρασμο ΣΥΝ εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το Brexit, επειδή λοιπόν δεν υπευλήθησαν αυτέ τι αντιρρήσει, θεωρείται ότι ενεκρίθησαν αυτές, οι, αυτή, ενεκρίθη αυτή η, ε, το σχέδιο έκθεση με βάση το άρθρο 50 παράγραφος 2 του ε, εσωτερικού κανονισμού. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το κείμενο και θεωρώ ότι θα εγκριθεί στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικά μέτρα για τον προπολογισμό του 2020. Όσον αφορά τον προπολογισμό αυτό, το έγγραφο εργασίας για αυτά τα PPPA θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 7 Μαρτίου και θα αναφέρει τις προτεραιότητες της κυρίας Χολμάρη που είναι η κυρία εισηγήτρια του Κοινοβουλίου. Κατόπιν οι Επιτροπές θα λάβουν περισσότερο ενημέρωση για τις προθεσμίες και τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβληθούν αυτές οι ενέργειες για μια προπαρασκευαστική αξιολόγηση. Θα ενημερωθείτε. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα ε, οργανώσει μία συνεδρίαση ενημέρωσης για τη διαδικασία προϋπολογισμού για το 2020 για, στις 8 Μαρτίου λοιπόν για τους συναδέλφους και τους ε, υπαλλήλους. Θα ενημερωθείτε για το χώρο και την ακριβή ώρα. Επίσης, σας είπα με mail ότι αμέσως μετά τις ψηφοφορίες θέλουμε να κάνουμε μια οικογενειακή φωτογραφία της Επιτροπής μας. Σας παρακαλώ να μην ε, τρέξετε να φύγετε όλοι μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, αλλά να μείνετε εδώ για να κάνουμε αυτή τη φωτογραφία. Η γραμματεία μας απέστειλε μάλλον η γραμματεία μας θα προετοιμάσει ένα φυλάδιο για τις εργασίες της Επιτροπής μας τα τελευταία πενταετία θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει και μία φωτογραφία και γι' αυτό σας παρακαλώ να μείνετε όλοι για να είστε σε αυτή τη φωτογραφία αυτά για τις ανακοινώσεις μου ψηφοφορίες λοιπόν έχουμε δύο σημαντικές εκθέσεις σήμερα για τις οποίες πρέπει να ψηφίσουμε και να ξεκινήσουμε σχέδιο έκθεσης για τον έρασμο που είναι το πρόγραμμα της Ένωσης για τη γενική και επαγγελματική κατάρτιση, την νεότητα και τον αθλητισμό. Να ρωτήσω το συνάδελφο αν θέλει το λόγο όχι. Ωραία. Πάμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Έχετε όλοι τις καρτούλες σας. Τις έχετε βάλει στο μηχάνημα. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 1. 84 και 85 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνονται. Α, και 86 και 87 ήταν ίδιες. Ωραία. Έμπλε 1. Συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι. Έμπλε 56, όχι. Συμβαστική 1-1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. εγκρινεται εγκρίνεται. Συμβαστική 1-2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1-3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2-1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2-2 στη σελίδα 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 2-3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 263 υπέρ. Στη σελίδα 28. 263. Α, όχι, σελίδα 29 καλύτερα. Σελίδα 29. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλά, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 9-18. 2-49. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 168 υπέρ κατά αποχές. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω τι γίνεται εκεί πέρα, παρακαλώ. Είναι εδώ η κάμερα μπροστά μου. Υπέρ, λέω. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία 13 υπέρ 13 κατά. Λοιπόν, συμβαστική 2-4 υπέρ. Κατά άποχες, δεκτή. Συμβαστική 3-1 υπέρ. Κατά άποχες, δεκτή. Συμβαστική 3-2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβαστική 3-3 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4-1 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4-2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4-3 4-3 λοιπόν, υπέρ. Κατά. αποχε δεκτη Δεκτή. Συμβαστική 5-1 υπέρ. κατα αποχε Αποχές. Δεκτή. 5-2 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, είναι ονομαστική ψηφοφορία. Η 5-2 είναι ονομαστική, άρχεται. Πέρας. 17-11. Οπότε καταπίπτει η 5-2α συμβαστική. Και περνάμε στην συμβαστική 5-3. Διαδικαστικό. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Υπά, έχουμε ένα λάθος ε, στον ε, κατάλογο ψηφοφοριών μας. Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία παρακαλώ. Όχι βέβαια, κανονικά. Μόνο αν δεν υπάρχει αντίρρηση, αν συμφωνούν όλοι. Ε, αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για να επανελθεί η ψηφοφορία για την 5-2, Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, λοιπόν επανερχόμεθα. Έχουμε δύο εναλλακτικού συμβιβασμού για το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 20, 25. Ε, Πρώτη δυνατότητα. Η συμβαστική του εισηγητή. Και η άλλη είναι η συμβαστική σοσιαλιστών Αλτεγκούε και Πρασίνων. Λοιπόν, Πρώτα να ψηφίσουμε την συμβαστική πρόταση 5-2, τη συμβαστική δηλαδή του εισηγητή και μάλιστα ονομαστικά. Άρχεται. Πέρας. Λοιπόν, απορρίπτεται με 9-20. Όντως κάποιο λάθος υπήρχε κάπου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και εγώ το πρόσεξα, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να σχολιάσω. Να περάσουμε τώρα στη συμβαστική 52α, επίσης ονομαστική, η οποία και άρχεται. Μάλιστα. Πέρας. Α, δεκτή. Δεκτή με ευρία πλειοψηφία 21, 21 ψήφι με 7. Λοιπόν, Τότε πάμε στο 5-3 λοιπόν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 6-1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 6-2. Είναι πολύ αργότερα παρακάτω. 6-2. Τη βρήκατε όλοι. Στη σελίδα 78, τώρα στη δική μου λοιπόν των σοσιαλιστών είναι στην 78, τώρα στον άλλον πολιτικό ομάδο δεν ξέρω. Συμβαστική 6-2. Τη βρήκατε όλοι. Οπότε ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή 6-3 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές δεκτή οπότε έχουμε την τροπολογία 2.72 2.72 Τη βρήκατε όλοι Ωραία, ποιος είναι υπέρ Κατά Αποχές, απορρίπτεται Συμβαστική 7-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 7-2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7-3. Στην επόμενη σελίδα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έμπλ 11 υπέρ. Κατά Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 8-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8-2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9-2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή budget 22 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε Budget 22 άρχεται στη σελίδα 101 Budget 22. Πέρας. Δεκτή 21 8. Συμβαστική 12. 12 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11. Όχι, συγγνώμη. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Α, α, είπα 15. Α, είπα το όπα το 15. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι, δεν χρειάζεται δύο φορές. Τελική ψηφοφορία, που είναι τρεις τελικές ψηφοφορίες. Όλες ονομαστικές. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε για τις τροποποιήσεις του σχεδίου νομοθετικής πρότασης. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Δεκτή 28 υπέρ και μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια. Τώρα ψηφίζουμε δεύτερη ψηφοφορία. Ονομαστική. Η συμβαστική 16. Ψηφίζουμε την συμβαστική 16 που είναι τροποποίηση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή τα ψηφί, 29 ψήφοι υπέρ. Και τώρα τελική ψηφοφορία και των δύο κειμένων από κοινού άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται με 28 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά. Σχεδόν παμψηφί. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Και βεβαίως επίσης τον ευχαριστούμε γιατί μας διευκόλυνε τη ζωή ιδιαίτερα με τις πολλές συμβαστικές και συγχαίρουμε λοιπόν και τους κοιόδης που έτσι πραγματικά απλούστευσαν την κατάσταση γιατί αν έπρεπε να ψηφίσουμε 100 σελίδες τροπολογίες θα είχαμε βαρεθεί ιδιαίτερα και θα ήταν και πολύ περίπλοκο και νομίζω ότι συνολικά είναι καλό το κείμενο το οποίο εγκρίναμε. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Συμβούλιο για να βρούμε τις σωστές λύσεις. Συγχαίρουμε λοιπόν ολόθερμα τους σκιώδεις και τον εισηγητή και φυσικά και τη γραμματεία μας, όλους τους συνεργάτες μας και των δύο φίλων οι οποίοι βοήθησαν τόσο πολύ, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα τόσο καλό κείμενο τώρα. Ακολουθεί η έγκριση σχεδίου εκθέσεως για, το, για την δημιουργική Ευρώπη με εισηγήτρια την κυρία Σίλβια Κώστα. Σίλβια, έχεις τον λόγο. Απλώς να ευχαριστήσω θερμά τους χειώδεις ε, εισηγητές, τους συναδέλφους από όλες τις ομάδες για την ε, συνεργασία και ιδιαίτερες ευχαριστήσεις προς τη γραμματεία, στην Γκόσα Λούκα ειδικά, στην κόσα και στο Λούκα μάλλον, γιατί με στήριξαν ιδιαίτερα και μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η επόμενη θητεία, πώς να το πω, θα ακολουθήσει αυτή την ε, αφετηρία για όλα τα αιτήματα προς τον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ Σίλβια. Να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία και αρχίζουμε με την συμβαστική 1. Παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές προτιμώ να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 28 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 14 υπέρ 11 κατά. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 32 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει πέρας απορρίπτεται 15 ψήφι κατά 14 υπέρ 34 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι και αυτή απορρίπτεται αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε στις 34 λοιπόν ηλεκτρονικά πέρας απερίφθη 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 ε, τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 341, 340 και 339 που είναι ταυτόσιμες, όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 347 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 348 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές προτιμώ να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 43 λέει η πρόεδρος 44 διορθώνει τώρα 44 λοιπόν 44 πέρας με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, μεγάλο άλμα, συμβαστική 81, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή. 406, τροπολογία 406, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Budget 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 408 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 409 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 410 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 412 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 413 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 414 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε 414 Τέλος, πρόκειται περί ισοψηφίας, απορρίπτεται. Παρατήρησε χωρίς μικρόφωνο. Νομίζω ότι μια ε, βουλευτής λέει ότι δεν πάτησε καλά το κουμπί. Α, δεν πρόλαβα να ψηφίσω. Συγγνώμη. Εγώ ήθελα όμως να υπερψηφίσω. Να με συγχωρείτε. Πού είχαμε μείνει, λέει η πρόεδρος. Νομίζω μπορούμε να δεχτούμε εφόσον δεν λειτουργήσε καλά το μηχάνημα, λέει ο πρόεδρος. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μια στιγμή να καταλάβω, λέει η κυρία Κώστα. Για το 54, όχι μάλλον, συγγνώμη, το 414, α, λοιπόν, εγκρίνεται, 414 εγκρίνεται, διότι ήταν ισοψηφία 14-14, η Μικαέλα υπερψήφισε, άλλα 15-14. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. 54 πάντοτε, 54. Προτιμώ να επαληθεύσουμε, να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο. Πέρας. Απορρίπτεται 18 κατά 11 υπέρ. 415 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 416 και 17 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτονται. 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 419 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 423 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 422 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 428 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 429 υπέρ. Κατά αποχές προτιμώ να κάνουμε ηλεκτρονική παρήθευση. 429 τέλος 18 ψήφι υπέρ 11 κατά 430 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 433 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 434 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 αυτή έχει αποσυρθεί Προφορική τροπολογία για την 438 τώρα της κυρίας Κώστα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 442 και 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 444 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 445 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 448 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 449 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 450 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, εγκρίνεται διορθώνει πρόεδρο. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Την ψηφίσαμε ήδη αυτήν. Με συγχωρείτε, λέει πρόεδρο. Νομίζω ότι ε, ε, δεν πρόλαβα καν κοιτάξω καλά και ξεφώνησα ήδη. Καλά, έστω. Για τους τύπους να ξαναψηφίσουμε 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 462 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Καλώς λοιπόν. Κάνουμε επαλήθευση. Πέρας. Η πράσινη ομάδα των πρασίνων έχει μία ψήφο παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει να αφαιρέσει κάποιο την κάρτα του. Τώρα λοιπόν ναι, εντάξει. Πέρας. Ψήφι 17 υπέρ, 11 κατά. 463 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Έχει καλώς. 69 ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος. 18 ψήφι υπέρ, 11 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Budget 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 470 υπέρ. Όχι, 471 λέει η πρόεδρος. Υπέρ. 471 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός 471 τέλος ψήφι 21 υπέρ 8 κατά τα χέρια σας δεν τα είχατε σηκώσει καλά 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 475 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 476 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αν θέλετε παρήθευση. 74. Ηλεκτρονική παρήθευση. Πέρας απορρίπτεται ψήφι 15 κατά, 14 υπέρ. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολύ μικρή διαφορά. Ας ευπαληθεύσουμε και εδώ. Τέλος. 14 ψήφι κατά 9 υπέρ. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 480 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση πάλι 77 τέλος 12 κατά 11 υπέρ απορρίπτεται 481 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 488 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 489 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Α, 82, 82 διορθώνει αμέσως. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 509 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Καλώς λοιπόν, επαληθεύουμε ηλεκτρονικώς την 83. Τέλος. 18 υπέρ, 10 κατά. 84 υπέρ, κατά. Αποχές. Κανένα χέρι σχεδόν δεν βλέπω να σηκώνεται. Επαλήθευση λοιπόν, 84. Τέλος, 18 προς 10 εγκρίνεται. Βλέπω σιγά σιγά να κουράζεστε. 85 υπέρ, κατά Αποχές. Πάλι επαλήθευση. 85. Πέρα τη ψηφοφορία, σαφή έγκριση. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά Αποχές. εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 517 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 518 υπέρ. Κατά. Αποχές. Χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση εδώ. 518. ισοψηφία. 14 προς 14, άρα απορρίπτεται. 87 υπέρ. 87 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 519 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 520 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ομοίως. Συμβαστική 47 υπέρ. Δεν έχει πει υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 523 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 524 υπέρ. 524 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση 524. Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 525 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 526 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 527 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές προτιμώ να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο Υπαριθμόν 90 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψήφι 13 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται Συμβαστική 49 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 51 έτσι λέει η πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 541 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 542 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 544 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 543 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 547 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 548 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 549 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 554 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 557 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 558 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 559 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 567 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 500 όχι, διορθώνει η πρόεδρος. Συμβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 575 υπέρ κατά αποχές. Εδώ χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. 575 είναι ο αριθμός της τροπολογίας που επαληθεύεται. 575. 575. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Συμβαστική 84 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε, η 7. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση 151. Πέρας. Ψήφι 16 κατά 13 υπέρ. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές πρότυπο να επαληθεύσουμε Υπαριθμόν 9 πέρας απορρίπτεται 15 κατά 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 και 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται προτιμώ να επαληθεύσουμε 160 πέρας πράγματι εγκρίνεται Συμβαστική 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Προτιμώ να επαληθεύσουμε για να είμαστε πιο σίγουρες. Πέρας. Α, απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός 196 πέρας απόρριψη 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Budget 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση 203. Πέρας. Απορρίπτεται 17 κατά 12 υπέρ. Συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 75 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικός τέλος ισοψηφία 14 προς 14 απορρίπτεται 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 και 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές προτιμώ να επαληθεύσουμε 223 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 231 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά αποχές σαν να μην ψήφισε το Λαϊκό Κόμμα. 251, ξαναλέω. Επαλήθευση όμως τώρα. Τέλος της επαληθεύσεως ψήφι 21 υπέρ, 3 κατά. Και 5 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. 252 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 254 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, ακολουθεί η τελική ψηφοφορία η οποία γίνεται ονομαστικά. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν. Τέλος. Ψήφι 28 υπέρ, καμία κατά και μία αποχή. Άρα, ομόφωνη έγκριση, συγχαρητήρια, θερμότατα. Σίλβια, μεγάλες ευχαριστίες επίσης στους ε, συνεισηγητές, την γραμματεία, και όλες και όλους τους συνεργάτες που με την προσπάθειά τους συνέβαλαν ώστε να έχουμε μια στέρεα κοινοβουλευτική θέση με την οποία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Συνεχίζει η πρόεδρος Κάμερ Θα προχωρήσουμε τώρα στην λήψη της φωτογραφίας. Θα ήθελα παρακαλώ πρώτα όλοι οι βουλευτές οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να συγκεντρωθείτε εδώ μπροστά και μετά θα ακολουθήσει μια δεύτερη φωτογραφία όπου θα συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτες και της γραμματείας και των πολιτικών ομάδων.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 Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα περνάμε στο σημείο 6 της ε, σημερινής μας συνεδρίασης. Είναι λοιπόν θέμα μίας μελέτης που παραγγείλαμε και την οποία ε, διεκπαιρέωσε και παρακολούθησε το τμήμα πολιτικής Β για την ε, πρόορια κατάληψη των σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και την προηγούμενη φορά έχουμε τα προσωρινά αποτελέσματα της μελέτης και πρώτον τι γίνεται στα κράτη-μέλη όσον αφορά το θέμα αυτό και αν υπάρχουν θετικά υποδείγματα πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πρόορη διακοπή σπουδών στην Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για μια ενημέρωση της προηγούμενης μελέτης που ήταν από το 2011 ε, αντιμετωπίζει τα, τις κυριότερες εξελίξεις ε, και τα αίτια του προβλήματος από τότε που υπήρχαν συστάσεις του Συμβουλίου 2011 για τη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος και πώς θα αναπτύξουν πολιτικές πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Η μελέτη είδε τη σχέση μεταξύ διακοπής ε, των σπουδών και των δημοσίων δαπανών και ε, υποβάλλει συστάσεις για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος να καλωσορίσω την κυρία Φαντενγκράφ από τον οργανισμό Παντία. Θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα για 10 λεπτά και κατόπιν θα έχουμε μία διαδικασία έρωτα απαντήσεων. Πριν σας δώσω το λόγο, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε εδώ 10 σπουδαστές από το γαλλικό νομό του Γκαρόν Κάνουμε μια σύγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον οργανισμό Καναδάς και Μπέκ Ευρώπη για τη συνεργασία που μπορούμε να έχουμε με τον Καναδά από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Είμαστε σε πολύ στενές σχέσεις πολιτιστικά με τον Καναδά, ιδιαίτερα για το γαλλόφωνο τμήμα του Καναδά. Γι' αυτό σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή μας και σας εύχομαι μία όμορφη και ενδιαφέρουσα παραμονή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι για την παρουσία σας. Και τώρα, κυρία Φάντερ Γκράφ, παρακαλώ, παρουσιάστε τη μελέτη. Χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να μπω απευθεία ε, στο ψητό, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Λοιπόν, ε, η θαυμάσια μελέτη μας ε, ήταν μια ενημέρωση της μελέτης του 2011 που είχε παραγγείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι και μετά θα σας πω και τα συμπεράσματα. Η μελέτη αυτή, όπως λέγεται, είναι μια ενημέρωση της μελέτης του 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν μια ε, μεγάλη διάσταση μελέτης, πολύ ενημερωτική και τώρα κάνουμε μια ενημέρωση για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Έγινε στα πλαίσια των συστάσεων του Συμβουλίου του 2011 για την πολιτική για το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη εκλήθησαν να εξετάσουν τα αίτια και του παράγοντε που προκαλούν το φαινόμενο αυτό, να ανταλλάξουν καλέ πρακτικέ και να αντιμετωπίσουν το θέμα. Και ε, να υπάρξει μια συνολική στρατηγική για το θέμα αυτό. Ποιοι είναι οι δικοί μα στόχοι. Θέλουμε να ενημερώσουμε στατιστικά τι έχει συμβεί τα τελευταία 7 χρόνια, να δούμε τι έχει αλλάξει, να δούμε τη σχέση μεταξύ δημοσίου δαπανών στην εκπαίδευση και διακοπή σπουδών και ποιε είναι οι μελλοντικέ τάσει και να κάνουμε και συστάσει. Πώς θα κάναμε αυτό. Κάναμε έρευνα γραφείου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεντεύξει σε έξι χώρε για έξι κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Λοιπόν, και πάλι στην ουσία, για να μιλάμε με βάση το ίδιο πλαίσιο, τι σημαίνει διακοπή των σπουδών είναι νέα άτομα μεταξύ 18 και 24 που δεν έχουν πάρει παρά μόνο το χαμηλότερο επίπεδο τη δευτερεύουσα εκπαίδευση και που δεν λαμβάνουν αυτή τη στιγμή καμία εκπαίδευση ή κατάρτιση. Στους 28 ο μέσο όρο είναι 16, 10,6 συγγνώμη, μεταξύ 11 και 17. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια μέση μείωση 2,8%. Πολλέ χώρε επέτυχαν του στόχου του, του εθνικού στόχου για τη μείωση του φαινομένου. 14 χώρες συγκεκριμένα και πολλές άλλες τον προσεγγίζουν το στόχο τους. Η καλύτερη είναι η Πορτογαλία, όπου μειώθηκε κατά 10,4% μεταξύ 11 και 17 το φαινόμενο, η Ισπανία 8%, η Ελλάδα και η Ιρλανδία επίση τα πάνε καλά. Τώρα οι βραδιπορούντες, Σλοβακία, όπου είχαμε αύξηση κατά 4,2% και στην Τσεχία και μας εξέπληξε η Σουηδία που υπήρξε μια μικρή αύξηση του φαινομένου αυτού ενώ γενικά τα πάνε πολύ καλά. Δεύτερος στόχος, αίτια. Τρία κύρια αίτια. Πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι σπουδαστές, το κοινωνικο-οικονομικό τους περιβάλλον, ε, το οικογενειακό περιβάλλον, το κόστος, ε, οι, ο, εκεί που μένουν, αν είναι στην Ήπεθρο ή στη, σε πόλεις, οι φίλοι τους, το φίλο και η εθνότητα των ε, μαθητών και ιδίω πόσο έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές αυτοί. Συστημικοί τώρα παράγοντες. Έχει να κάνει με τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι ε, διαστάσεις του σχολείου, που βρίσκεται το σχολείο, οι εκπαιδευτικές πρακτικές και η ποιότητα των εκπαιδευτικών. Και τέλος, ε, το εθνικό πλαίσιο επίσης μπορεί να παίξει ρόλο. Η αγορά εργασίας, για παράδειγμα, η οικονομική κατάσταση, σημαντικοί παράγοντες, η πολιτική κατάσταση, και οι πολιτικές που έχουν οι κυβερνήσεις για την αγορά εργασίας, για την, για την εκπαίδευση και οι στάσεις της κοινωνίας. Και επίσης σε μικρότερο βαθμό η αντιμετώπιση των μειονοτήτων. Τώρα, το φαινόμενο αυτό είναι μια διαδικασία. Η διακοπή σπουδών είναι μια διαδικασία. Δηλαδή προκύπτει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Όλοι οι παράγοντες αυτοί αλληλοπιδρούν και αυξάνουν ή μειώνουν το ενδεχόμενο να καταλήψει ένα σπουδαστή τι σπουδέ του. Ένας μαθητής επίσης. Οι ίδιοι παράγοντες λοιπόν έχουν άλλο αποτέλεσμα ανάλογα με τις χώρες. Να μην το ξεχνάμε. Τι πολιτικές παρεμβάσεις ε, τώρα μπορούν να μειώσουν το φαινόμενο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για τη διακοπή σπουδών συνήθως αντιμετωπίζεται έμεσα μέσω των πολιτικών για την αγορά εργασία, την εκπαίδευση ή την κοινωνική ένταξη. Και τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι παρεμβάσεις πολιτικής. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επειδή είναι περίπλοκο φαινόμενο και οφείλεται σε πολλούς λόγους, πρέπει να υπάρξει συνολική προσέγγιση αν εξετάσουμε κατά κράτο, είναι δύσκολο να δούμε πώ μια συγκεκριμένη πολιτική παίζει ρόλο. Είναι δύσκολο να απομονώσει και να εξετάσει το αποτέλεσμα μια πολιτική. Γι' αυτό οι, μελέτες, ε, οι μελέτες ε, ε, αντικτύπου είναι δυσχερείς, αλλά παρόλα αυτά επιχειρούνται. Τρεις τύποι παρεμβάσεων μπορούν να γίνουν. Πρόληψη, παρέμβαση και επανένταξη ή αντιστάθμιση. Λοιπόν, πολιτικές πρόληψης για να μην ε, διακόπτουν λοιπόν οι σπουδαστές τις σπουδές τους. Πρέπει για παράδειγμα οι βαθμοί να μην διατηρούνται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί αυτό έχει αποτέλεσμα στην διάθεση των μαθητών να συνεχίσουν εξωσχολικές δραστηριότητες και μέτρα για να ενταχθούν ε, τα παιδιά των μεταναστών που μόλις έχουν φτάσει. Επίσης καλή προσχολική φροντίδα ε, ελκυστικές δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και περισσότερη ε, αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων εκπαίδευση, Να υπάρχουν, για παράδειγμα, επίσης ε, απουσιολόγια, να βλέπουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πόσοι εγκαταλείπουν και να υπάρχουν μέτρα θετικών διακρίσεων και πολιτικές για να μην απομονώνονται κάποιες κοινότητες. Παρεμβατικές πολιτικές τώρα. Για, εδώ πρέπει να δούμε τους φοιτητέ και τους σπουδαστέ καλύτερα που κινδυνεύουν να καταλήψουν την εκπαίδευση ή κατάρτιση. Είναι πιο ευάλωτοι. Πρέπει να καταρτίζονται ακριβώς οι εκπαιδευτικοί για να βοηθούν τους φοιτητέ, Ιδιαίτερα να τους βοηθούν γλωσσικά και ειδικευμένο προσωπικό για να ε, στηρίξει τους εκπαιδευτικούς για να αναγνωρίζουν τα προμηνύματα της εγκατάλειψης των σπουδών και η εκπαίδευση των ίδιων των ε, γονέων και κηδεμόνων. Και οι φοιτητέ ε, και σπουδαστέ που έχουν εγκαταλείψει την κατάρτιση και εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικέ επανένταξη και αντιστάθμιση. Να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα δεύτερη ευκαιρία που μπορεί να έχει διάφορε μορφέ. Εναλλακτικά μέτρα επίση. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν να επανενταχθούν οι σπουδαστέ που έχουν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό σύστημα. Γενικά λοιπόν, οι χώρες υιοθετούν ε, ένα σύνολο τέτοιων μέτρων προληπτικών παρέμβασης και επανένταξης. Είναι δύσκολο να δούμε τι αποτέλεσμα έχει αναχώρα ένα συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής. Τρίτος στόχος. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης, της, ε, των δημοσίων επενδύσεων στην εκπαίδευση και του φαινομένου. Εξετάσαμε τι ε, δαπάνε για την εκπαίδευση ω ποσοστό του ΑΕΠ των διαφόρων χωρών σε σχέση με το ποσοστό διακοπή σπουδών και αν έχει μειωθεί την τελευταία επταετία, δηλαδή την επταετία καλύτερα 11-17. Πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει γραμμική άμεση σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών δαπανών και διακοπής σπουδών. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, και την Ιρλανδία, που δαπανούν τα λιγότερα ενώ τα πάνε πολύ καλά στην μείωση του φαινομένου διακοπής. Και το αντίθετο είναι η Σουηδία, που τα πάνουν πάρα πολλά, αλλά είδαμε ότι αυξήθηκε ελαφρώς το φαινόμενο διακοπής σπουδών. Άρα, τι σημαίνει όλα αυτά για την Ελλάδα, για παράδειγμα. Πολύ, πολλές επενδύσεις στην εκπαίδευση είναι ιδιωτικές, όχι δημόσιες χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει σχέση, αλλά δεν είναι άμεση και γραμμική, είναι πιο περιπλοκή. Όπω είπα, χρειάζεται περαιτέρω εξέταση. Λοιπόν, στις συνεντεύξει διαπιστώσαμε ότι το θέμα δεν είναι πόσα, αλλά πώς θα δαπανά. Επειδή πολλά αίτια οδηγούν στη διακοπή. Άρα χρειάζεται συνδυασμό μέτρων για να αντιμετωπιστεί. Καλά, αυτό δεν είναι και τόσο πρωτότυπο. Αλλά εξαρτάται από τι προκλήσει και τα αίτια σε κάθε χώρα. Άρα χρειάζεται πιο εστιασμένη αντιμετώπιση, βλέποντα ποια είναι ακριβώ τα αίτια. Συστάσει τώρα. Βλέπετε εδώ μερικέ από τι κύριε συστάσει. και από τα, τις μελέτες που ε, εξετάσαμε και από τις συνεντεύξεις. Πρώτον λοιπόν να υπάρχει ένα μητρό απουσιών, απουσιολόγια. Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμήματων και υπηρεσιών. Να υπάρχουν συνολικές στρατηγικές. Ορισμένες χωρίς το κάνουν, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Να κοιτάξουμε σε τοπικό επίπεδο τις ανάγκες των ε, σπουδαστών και να είναι πιο προσβάσιμη η σχολική εκπαίδευση για τις ομάδες που ε, είναι πιο δύσκολο να ενταχθούν σε αυτήν. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Να βοηθήσουμε αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο. Σε σχολείο και σε εθνικό επίπεδο. Σχετίζεται με τις δύο προηγούμενες ε, συστάσεις. Και συστημικά περισσότερη εκπαίδευση και βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν πώς θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τους μαθητές από διαφορετικά, ε, διαφορετικής προέλευσης και σε επίπεδο ένωσης να υπάρξει ευαισθητοποίηση για τη διαθεσιμότητα πόρων ενωσιακών για να βοηθηθούν αυτές οι πολιτικές όπως το Ερασμό για παράδειγμα. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος Κάμερεβερτ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Είναι θετικό το νέο ότι από ό,τι φαίνεται σε πολλές χώρες μέλη έχει μειωθεί ο, ρυθμός, ο άριθμος καλύτερα των προσώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες επιτυγχάνουν. Κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προβάλει τον στόχο του 10%. Φαίνεται πως αρκετές χώρες μέλη το επιτυγχάνουν ή πάντω βρίσκονται σε καλό δρόμο για να το επιτύχουν. Προσωπικά, εγώ βρίσκω πάντοτε το 10% υπερβολικά υψηλό και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε ή δυνατόν να δώσουμε σε κάθε παιδί πιθανότητε, δυνατότητε, να αυτονομηθεί στη ζωή του μέσω μια στέρεα παιδείας. Νομίζω λοιπόν ότι όντω χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειε. Υπάρχουν και ορισμένα α, πορίσματα τα οποία εκπλήσουν, ίσω μπορείτε να τα σχολιάσετε περισσότερο, ειδικό στη Σουηδία που ε, συνήθως ε, προβάλλεται ως πρότυπο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φαίνεται ε, λοιπόν ότι εκεί ο αριθμός των προσώπων που καταλήπουν το σχολείο αυξάνεται στο λίγο. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, κάποια αιτιολόγηση, να μας την πείτε. Υπάρχουν όμως και θετικά παραδείγματα εκεί όπου δεν τα περιμέναμε. Ελλάδα για παράδειγμα, Πορτογαλία επίσης, όπου γνωρίζουμε ότι οι χώρες αυτές, ιδίως ό,τι αφορά τους ε, δημόσιους προϋπολογισμούς τους δεν είναι πολύ ε, ας πούμε ευπαρκής. Γι' αυτό το ερώτημα είναι πόσο, πόσα χρήματα δαπανώνται, επενδύονται στην παιδεία και πάντως όχι γραμμικά για να δούμε σε ποια αναλογία βρίσκονται οι επενδύσεις αυτές με τους αριθμούς των ε, μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, μπορούμε να προχωρήσουμε ε, σε συζήτηση. Και πρώτη, κυρία Βερχάιεν, επανέρχομαι σε ένα θέμα. Οι top performer, όπως είπατε, είναι Πορτογαλία, Ισπανία, ε, Ιρλανδία. Δηλαδή, κατά παράδοξο τρόπο, οι χώρες οι οποίες πέρασαν από τη βαθύτερη οικονομική κρίση. Και όπου βέβαια εκεί υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν και τα κονδύλια της εγγύησης ε, για τους νέους. Η μείωση τώρα των χρηματοδοτήσεων ε, για... Βρίσκονται τα κονδύλια της εγγύησης ε, των νέων σε άμεση σχέση με την μείωση των προσώπημα για τα το σχολείο. Κάτι το οποίο δεν συνέβη, α πούμε, στη Σουηδία. Δεν πήγαν το ίδια κονδύλια στην Σουηδία, για παράδειγμα. Μπορείτε να πείτε κάτι σχετικά. Και επίση, άλλη ερώτηση. Είπατε ότι έγιναν έξι μόνο περιπτώσει. συζητήσατε. Είναι αλήθεια αυτό ή πόσε χώρε εν πάση περιπτώσει ήταν. Γιατί στη διαφάνεια 3 βλέπω ήδη να αναφέρονται 7 χώρε. Ποιες σε ποιες χώρες στόχευσε λοιπόν η έρευνα. Επίσης η διαφορά ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα παίζει κάποιο ρόλο όπως για παράδειγμα η δυτή ε, παιδεία που έχουμε εμείς στην ε, Γερμανία που έχει και επαγγελματική κατάρτιση ε, παίζουν εκεί κάποιο ρόλο για, τους, για το early school living. Ωραία, θα κάνουμε όπως κάνουμε συνήθως, δηλαδή εν είδη αντισφαιρίσως. Γι' αυτό θα δώσω απέσως το λόγο στην κυρία Ντεγκράφ για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα αρχίσω με το πρώτο για την ε, εγγύηση για τους νέους. Ρίξαμε μια ματιά συνολική ε, στην χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν μπήκαμε σε πολλές λεπτομέρειες. Είναι περισσότερο μια μελέτη ενημερωτική, update δηλαδή, και εξετάσαμε τις εθνικές πολιτικές και τα προγράμματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την Youth Guarantee δεν μπορώ δυστυχώς να δώσω πολλές πληροφορίες. Ίσως είναι μια χρήσιμη προσθήκη στην μελέτη που θα πρέπει να γίνει ακόμη βέβαια. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των χωρών μελών, πράγματι εξετάσαμε έξι. Σύμφωνα με τη γεωγραφική τους τοποθέτηση, πόσο καλά τα κατάφεραν στην προσπάθεια να μειώσουν την ε, πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου και υπήρχε και ένα κριτήριο ακόμη άνε ναι, ο αριθμός του πληθυσμού, το μέγεθος του πληθυσμού. Διότι παίζει ρόλο εκεί για το πόσο συγκεντρώνονται τα κονδύλια ε, υπέρ της παιδείας. Πόσο, ποια είναι η αναλογία δηλαδή και αν, είναι, αν υπάρχουν ε, μεγάλε μεγάλες εκτάσεις υπαίθρου κλπ. Άρα παίζει και η γεωγραφία των χωρών εκεί ένα ρόλο. Εν τέλει καταλήξαμε, όπως είπα, σε έξι χώρες μέλη. Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβακία. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πιέρ, που μου υπενθύμησε στην Σλοβακία. Επιλέξαμε επίτηδε να υπάρχει ένα μείγμα διαφορετικών χωρών και όντως μας εξέπληξε και μας ε, το χώρισμα για την ε, Σουηδία, ενώ άλλε χώρε όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα αντιμετώπισαν βαριά κρίση. Έχει πολύ ενδιαφέρον Ιρλανδία και Ελλάδα βρήκαμε πολύ υψηλότερο αριθμό στοχευμένων πολιτικών. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία, σε τοπικές κοινότητες, με συμμετοχή και των τοπικών κοινοτήτων και των σχολείων, ώστε να εξασφαλίσουν μια πιο συνολική προσέγγιση για την στήριξη των ε, παιδιών εκείνων που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Και με πολιτικές οι οποίες στόχευσαν ειδικά σχολεία σε φτωχές περιοχές ώστε να τους προσφέρουν ιδιαίτερους πόρους και στην Ελλάδα με θέματα μετανάστευσης τα οποία αντιμετωπίζουν είδαμε πολλές πολιτικές που στόχευαν στην ένταξη των παιδιών των μεταναστών και προσφύγων Εκεί προσφέρεται και ειδική εκπαίδευση για να εκπάθουν την ε, γλώσσα της χώρας. Στην Σουηδία είδαμε ότι αυτό δεν σημαίνει τόσο πολύ. Είδαμε μια ένα αυξανόμενο διαχωρισμό των παιδιών, παιδιών δηλαδή με μεταναστευτικό ε, ιστορικό, από τα παιδιά που δεν έχουν τέτοιο. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μάλλον συστήματα, δεν ήταν τόσο πολύ το κριτήριο επιλογής των χωρών, παραμείναμε στα κριτήρια που σας εξήγησα ώστε να έχουμε μια ευρύτερη επισκόπηση. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Μαρή Τερέζ Χιμένες, ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την... Ε, σας ευχαριστώ για την εργασία σας. Τι γίνεται με τους μαθητές μας, ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχουν διακρίσεις, βοηθάμε, προσέχουμε ιδιαίτερα ε, και για τις γυναίκες, ιδίως για τα κορίτσια. Αλλά βλέπουμε ότι η αποτυχία στο σχολείο συνήθως αφορά τα αγόρια. Τους εφήβους. Τι κάνετε γι' αυτό. Μήπως αντιδράτε υπερβολικά αργά επειδή εμεί λέμε ότι κυρίω πρέπει να ασχολούμεθα με τα κορίτσια, επειδή οι γυναίκε υφίστανται διακρίσει, αλλά δεν κάνουμε κάτι, θα γίνει πολύ σοβαρό το θέμα. Και δεύτερο, τι γίνεται στην Ισπανία, Μήπω έχει περισσότερε πληροφορίε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φαντεγράφ. Ευχαριστώ. Για να δούμε λίγο. Για τα ποσοστά εγκατάλειψης που αναφέρατε. Οι πολιτικές είχαν λάβει υπόψη τα ποσοστά εγκατάλειψη και ήταν ανάλογα με κατηγορίες και ανάλογα με τις χώρες. Η Ισπανία δεν ήταν από τις χώρες που μελετήσαμε. Είδαμε αν υπάρχει ποσοστό μείωση και στην Ισπανία τα πράγματα δεν ήταν πολύ κακά τα αποτελέσματα. 8% ε, μόνο. Τώρα για την ισότητα των φίλων στην εκπαίδευση. Δύσκολη ερώτηση. Πού να την απαντήσω. Στην ηλικία που είναι μεγαλύτερη η απειλή, το κίνδυνος για εγκατάλειψη, Όντω όντως οι περισσότεροι που φεύγουν είναι αγόρια. Ε, Έχουμε δηλαδή μια τάση να επικεντρώνουμε την ισότητα των φύλων στα κορίτσια, αλλά στην εγκατάλειψη βασικά αυτοί που φεύγουν από το σχολείο είναι τα αγόρια. Έχουν λιγότερη δυσκολία, ευκολία να συγκεντρωθούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διάφορε δυσκολίε συγκέντρωση τη προσοχή και ούτω καθεξής. Δεν το λέω εναντίον των αγοριών. Δεν έχω τίποτα μαζί του, αλλά ε, η πολιτικέ που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φίλου και στο επίπεδο τη εκπαίδευση θα είναι σημαντικό. Διότι τα αγόρια σε αυτή την ε, ηλικία δυσκολεύονται περισσότερο από τα κορίτσια. vielen Bild. Ευχαριστούμε κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία μου. Αναφερθήκατε στη Σουηδία που παρά τις εκπαιδευτικές δαπάνες που είναι από τις πλέον μεγάλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον ΑΕΠ βλέπουμε να εγκαταλείπουν το σχολείο οι μαθητές. Πιστεύετε ότι μεταξύ των δημόσιων δαπανών ε, και της σχολικής αποτυχίας να μην υπάρχει ένας σαφής δεσμός. Μετά βλέπουμε και σχέση με τη μετανάστευση και την πτώση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων. Διότι τα παιδιά των μεταναστών ή από προέλευση μεταναστευτική έχουν περισσότερο κίνδυνο. Έχετε μελετήσει τους συγκεκριμένου λόγους για την κατάσταση της Σουηδίας. Έχει καμιά σχέση η μετανάστευση ε, με όσα συμβαίνουν για την περίοδο που μελετήσατε. Και ε, ε, η συζήτηση που κλονίζει τον κόσμο τη εκπαίδευση συνοψίζεται στα εξή. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την εγκατάλειψη του σχολείου πρώτα ή να διαφυλαχθούν τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα. Στη Γαλλία, λόγου χάρη, το επίπεδο του μπακ του απολυτηρίου έχει γνωρίσει κάθε επιπτώση. 80% ε, επιτυχία έχουμε, την έχουμε διασφαλίσει, αλλά στην ουσία αυτό το απολυτήριο έχει χάσει πια την αξία του και δεν μπορεί πλέον κανεί με αυτό να βρει μια δουλειά. Άρα, η ε, ε, μείωση του επίπεδου, του εκπαιδευτικού επίπεδου, παρατηρείται παντού στην Ευρώπη, στην, ε, στο Βέλγιο, α πούμε, το ΣΕΜ. Εδώ, πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η καταπολέμηση τη εγκατάλειψη δεν θα μα οδηγήσει σε μία ισοπαίδωση των ακαδημαϊκών προτύπων. Ευχαριστούμε, κυρία Φαντεγκράφ. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Πρώτα για τη Σουηδία. Όντω, μελετήσαμε τη Σουηδία και η κατάσταση όπως και εσείς την σκιαγραφίσατε υπάρχουν ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Και βάσει των ε, επιστημονικών στοιχείων που μελετήσαμε, μπορεί κανεί να διαρρέσει τα πράγματα σε Σουηδούς και με Σουηδού. Μπορεί να είναι μετανάστες, μπορεί να έχουν ε, άλλους λόγους, που δεν είναι Σουηδοί. Αλλά τα πράγματα στη χώρα είναι γύλα. Σίγουρα υπάρχει σχέση μεταξύ δημόσιων δαπανών και σχολικής αποτυχίας, αλλά δεν είναι γραμμική η σχέση, δεν είναι απευθείας διασύνδεση αυτή που γίνεται. Τώρα για την πρόορα εγκατάλειψη του σχολείου, την υποβάθμιση των πτυχίων και των σχολικών διπλωμάτων, αυτό έχει να κάνει και με τα θέματα της πολιτικής εργασίας και κοιτάξαμε σε διάφορες χώρες τι γίνεται και πώς μπορούν να προσαρμόσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και αυτές που διδάσκονται και μαθαίνουν οι μαθητές μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό που βλέπουμε και αυτό προκύπτει και από άλλες μελέτες που εκπονήσαμε πρέπει να ξανασχεδιάσουμε τις δεξιότητες που προτείνουμε και διαθέτουμε στους μαθητές προς διδασκαλία. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής. πρέπει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις. να μάθουν και να καταλάβουν τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις. τι θέλουν να μάθουν οι μαθητές. Και αυτό πρέπει να γίνει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Προσωπικός, και αυτή είναι τελείως προσωπική άποψη, το υπογραμμίζω, θα έτεινα περισσότερο να καταπολεμήσω την σχολική υποτυχία, γιατί έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή ενό ανθρώπου. Από την υγεία του, την ψυχική του υγεία, μέχρι τι κοινωνικομικέ συνθήκε που ζει, την ψυχολογία. Είναι λοιπόν σημαντικό να το ερευνήσουμε και από μια διαφορετική σκοπιά σίγουρα και τι δεξιότητε σε σχέση με τι απαιτήσει τη αγορά εργασία. Αλλά υπάρχουν μελέτε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα μπορούσα να σα δώσω και κάποιε βιβλιογραφικέ αναφορέ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης βαθμίδας, εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντική για να μπορεί κανείς να πάει καλά στη ζωή του. Στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Είναι προϋπόθεση, έλεγα. Αν πρέπει να κάνουν κάτι τα κράτη-μέλη και η Ένωση, πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε τους στόχους. Θέσαμε ως στόχο το 10% αυτό να υπάρχει μόνο εγκατάλειψη σπουδών. Για να τον επιτύχουμε αυτό το στόχο έχουμε διάφορα μέσα. Έχουμε τον έρασμο συν συν, ε, το μέσο για την εγγύηση για την νεότητα και νομίζω ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας της χρήσης τους είναι διαφορετικός. Πρέπει να στηρίξει περισσότερο ενώ στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Είδαμε έξι χώρες εδώ πέρα. Ορισμένε ορισμένες τα πήγανε καλά, ενώ ορισμένες μείωσαν την παρέμβασή τους. Η Τσεχία είναι μεταξύ των κρατών όπου αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών και σπουδαστών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Είμαστε στο 5%. Δηλαδή λίγα παιδιά εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Λοιπόν, παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που έχουμε εδώ να μας πει εάν κατά την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων φροντίζουν τόσο ώστε να γίνεται καλύτερη ε, αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φάντερ Γκράφ. Ευχαριστώ για το σχολείο. Τι να συμφωνήσω για να είμαι ειλικρινής. Τι να σας πω. Πλάκα κάνω, αλλά... Πολύ δικαιούχοι αυτού του είδους των προγραμμάτων δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιες φορές. Και αν το γνωρίζουν, τα χρησιμοποιούν σαν κάτι επιπλέον. Και είμαι λίγο προκατηλημένη. Προέκυψε από τη μελέτη μας για το πρόγραμμα Erasmus In. Ίσως και η επικοινωνία και η προώθηση των προγραμμάτων αυτών δεν είναι σωστή. από την προοπτική των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Θα μπορούσαν και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και όλοι να σχεδιάσουν καλύτερα τα προγράμματα αυτά, δηλαδή την επικοινωνιακή του προβολή. Και δεν θα ήταν τόσο δύσκολο να προωθηθούν και να τα πουλήσουμε. Η διαδικασία υποβολή αιτήσεων ήταν τρομακτική για του περισσότερου χρήστε στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχεδιασμό και έχει του λόγου του. Ξέρουμε ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται έχουν συγκεκριμένου στόχου, δείκτε, αξιολογικού δείκτε κτλ. Και όλα αυτά που καταλάβουν τα ε, αρμόδια όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα αξιολογήσουν. Όμω για του δάσκαλου που πρέπει να συμπληρώσουν τι αιτήσει αυτέ είναι πολύ δύσκολα. Είναι περίπλοκα, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Πρέπει να επενδύσουν χρόνο. Και οι δάσκαλοι, όπω ξέρετε, ούτω ή άλλω είναι πιεσμένοι χρονικά. Τι να πρώτο κάνουν. Οπότε ο συσχετισμό αυτό μεταξύ των προγραμμάτων και των τελικών δικαιούχων, τέλο πάντων των πιθανών τελικών δικαιούχων, είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε καλύτερα. Να είναι η γλώσσα λίγο πιο εύληπτη. Να ασχολούνται οι δημοτικέ αρχέ, α πούμε, οι τοπικέ κυβερνήσει. Διότι θα έπρεπε να γνωρίζουν την ιδιαίτερη αξία των προγραμματών αυτών. Και θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ αυτό είναι το διαρκές μας αίτημα και ο διαρκής μας αγώνας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να απλουστευτούν τα πράγματα έτσι, κυρίως τα έντυπα αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις που να είναι κατανοητά και από τον απλό άνθρωπο. Να μην χρειάζεται να συμπληρώνει 50 σελίδες για να συμπληρώσει μια αίτηση. Τώρα, η Julie Ward, Ευχαριστώ πολύ. Ε, σημαντικό το θέμα. Διότι άπτεται τόσων πολλών πολιτικών τομέων. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπαίδευση. Έχει να κάνει με την αγορά εργασία. Θέματα βιωτικού ε, επίπεδου έχουν να κάνουν ε, με αυτό. Εγώ έχω εργαστεί με πολλούς νέους που έχουν περάσει από αυτές τις κοινωνικές δοκιμασίες. Ε, ξέρω νέους πολλούς που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Είχα μια ένωση καλλιτεχνών, ε, την οποία διευθυνά, η οποία πρότεινε ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ένα φάσμα υποστήριξης, ε, ειδών υποστήριξης ε, και εντός και εκτός σχολείου. Εάν δεν έχουμε εδώ μια σφαιρικότερη προσέγγιση, αν σκεφτούμε μόνο την εκπαίδευση και δεν σκεφτούμε το παιδί, το νέο σύνολο, την κοινότητα στην οποία ζει και να ρίξουμε ε, τα εμπόδια του και τα σύνορα μεταξύ του τι συμβαίνει εντός και εκτός σχολείου θα σφάλουμε. Οι νέοι μου φαίνεται ότι για να μάθουν, να διδαχθούν, να θέλουν, να επιθυμούν να είναι στο σχολείο, αυτό είναι άλλο θέμα. το, ζήτημα είναι να έχουν την επιθυμία να βρίσκονται στο σχολείο. Το κλίμα στα σχολεία, ποιο είναι, τα κοιτάξατε αυτά, είδατε ποιο, είναι το κλίμα στα σχολεία, η ατμόσφαιρα που επικρατεί στα ιδρύματα. Υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν ε, μαθητικά συμβούλια. Οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τι δικέ του ιδέες για το πώ θα έπρεπε να διευθύνεται το σχολείο, να είναι ένα ωραιότερο μέρο και καλύτερο μέρο για αυτούς. Αυτά είναι σημαντικά. Και στη δική μου τη χώρα έχουμε ένα βιογραφικό που γίνεται όλο ένα και πιο στενόμυαλο. Αυτό έχει ένα ε, όλο ένα και πιο ε, περιορισμένο κύκλο σπουδών. Αυτό ε, έχει να κάνει με πολλά θέματα και μαθήματα που έχουν ε, αφαιρεθεί από τον κύκλο σπουδών και δεν προσφέρονται στους νέους. Τα, ο αθλητισμός, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν έχουν απαραίτητο να κάνουν με το να κάθεται κανείς σε μια τάξη, να κοιτάει τον πίνακα και να μαθαίνει πράγματα απ' έξω για το τεστ και τις εξετάσεις που τον περιμένουν. Πρέπει τα πράγματα να τα δούμε λίγο σφαιρικότερα λοιπόν, όπου Εμεί θα πληρώσουμε το τίμημα αργότερα έτσι κι αλλιώ το οικονομικό κόστο των νέων που ε, δεν ε, μένουν στο σχολείο. Και ένα τελικό σχόλιο έχει να κάνει με τη χώρα σου, Πέτρα. Διότι έμαθα πρόσφατα ότι η Γερμανία, στη Γερμανία, η υπηρεσία για του νέου, η Jugendamt, είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά και υποστηρίζεται και από την κυβέρνηση. Εάν οι νέοι δεν έχουν καλές υπηρεσίες από αυτόν τον φορέα, μπορούν να υποβάλουν προσφυγή. Δηλαδή, υπηρεσία για την νεότητα μαζί με το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα μπορούσε να είναι μέρος της απάντησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φάνταγκραφ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και τα σχόλιά σας. Ενδιαφέροντα όσα έμαθα, καθώς έχετε και προσωπική εμπειρία φαντάζομαι ήταν ενδιαφέρουσα και σας και ικανοποιητική και για σας ως προς το κλίμα στα σχολεία σίγουρα παίζει ρόλο και κάνει διαφορά αυτά όμως είναι θέμα παρέμβασης στο επίπεδο του συστήματος και από την μελέτη ήταν δύσκολο να καταγράψουμε σε ποσοτικούς δείκτες τι κάνει την ατμόσφαιρα καλή σε, πολλά, σε πολλές συνεντεύξεις και λίματα και στοιχεία φαίνεται ότι οι δάσκαλοι είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Η υποστήριξη προς τους μαθητές ακούγεται καινοτοπία, αλλά είναι σημαντικά τα μαθητικά συμβούλια και προσφέρουν κάτι που σε πολλά σχολεία εύκολα το ξεχνάνε μελέτη δείχνει ότι έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζουμε συνήθω για να μείνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, κάπω να μπορούν να ταυτιστούν με τι δυσκολίε των διδασκόντων, με την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκαίρω. Για τι εξωσχολικέ δραστηριότητε, επίση πολύ σημαντικό, όλε αυτέ έχουν να κάνουν με το να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των μαθητών. Τα συμβούλια, ε, τα εξωσχολικά, ο αθλητισμό, εκφράσει μη ακαδημαϊκέ κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το αίσθημα του ανήκειν που μπορεί να δώσει και κίνητρα για να θέλει κανείς να μάθει, για τη μάθηση και για να είναι στο σχολείο. Οπότε ναι, ε, συμφωνώ. Τώρα για, τα, για την ύλη, για τα θέματα και τα μαθήματα που διδάσκονται. Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση και την βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα, κάποιοι σκέφτονται ας πούμε, ότι οι τέχνες και η δημιουργικότητα θα μπορούσε να είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σίγουρα υπάρχει μια τάση διακριτικής μεταχείρισης προς στιγμή. Αυτά είναι τα σχολεία μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λουίτζι Μόργανο. Ευχαριστώ. Θέλω από τη δική μου τη σκοπιά να ζητήσω μια διευκρίνηση. Ως Κοινοβούλιο και προσφάτω επαναλάβαμε την επιθυμία μας να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση των ε, πανεπιστημιακών διπλωμάτων, αν μη τι άλλο. Μιλάω δηλαδή για την ε, ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και το κ.ο.κ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αντικειμενικά διαφορέ στου κύκλου σπουδών σε διαφορετικέ χώρε. Όχι μόνο στι ε, παρόμοιε, αλλά και στι περιοχέ αναφορά που μελετήσατε κι εσεί στην μελέτη σα. Ένα πρόβλημα λοιπόν δεν νομίζω ότι βρέθηκε στο επίκεντρο τη προσοχή σα. Όχι ότι δεν θέλατε να το κάνετε, αλλά δεν μπορέσατε να το συμπεριλάβετε η σχέση μεταξύ των κύκλων σπουδών, των προγραμμάτων που προτείνονται στους μαθητές, δηλαδή το πόσο ζητούν ε, να καταβάλει κανείς προσπάθεια σε επίπεδο ε, των επιμέρους χωρών και της σχολικής εγκατάλειψης. Εδώ πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο στα γενεσιουργά αίτια, διότι δεν θα μπορούμε ούτε για την αγορά εργασίας να κάνουμε κάτι και το τρίτο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί θα είναι να μην έχουμε και συγκρίσιμα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Φάνταγ. ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρέπει να πω ως προς τις, τις απαιτήσει των κύκλων σπουδών, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τώρα σας μεταφράζω τις σκέψεις μου. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Το απαιτητικό είναι σχετικό. σε μια χώρα το ίδιο μάθημα μπορεί να το διδάσκουν πολύ διαφορετικά από την σε μια άλλη. Στη Φινλανδία, α πούμε, ήδη στο δημοτικό υπάρχουν καινοτόμε εκπαιδευτικέ ε, πρακτικέ. Οι μαθητέ δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα μαθήματα. Τέσσερι ώρε τη μέρα πάνε στο σχολείο και μετά εξερευνούν, α πούμε, τον κόσμο γύρω του. Αυτό καλλιεργεί την, ε, και οξύνει την περιέργεια, την φιλομάθεια. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι αυτό είναι απαιτητικό, διότι αναθέτει πολύ περισσότερες ευθύνες στους ίδιους τους μαθητές. Κάποιοι πραγματικά ανθίζουν και οριμάζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εγώ, ας πούμε, που είμαι πιο συνηθισμένη σε παραδοσιακά, ε, σε παραδοσιακούς κύκλους μαθημάτων και προγράμματα, θα μου φαίνονταν δύσκολο. Ε, το τι είναι απαιτητικό λοιπόν είναι διαφορετικό και παίζει σίγουρα ρόλο. Πάντως πάντοτε παίζει ρόλο και η ίδια ψυχολογική κατάσταση του μαθητή, η διάθεσή του για μάθηση που παίζει τον πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο του σχολείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης και τη δυνατότητα που μας δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις και εμείς οι ίδιοι έχουμε προχωρήσει σε αξιολόγηση της συστάσεως του 2011 και έχουμε συζητήσει και μαζί και θα συνεχίσουμε να συζητούμε και για όσους, με όσες και όσους ε, εξημών ε, επανέλθετε μετά τις ευρωεκλογές. Έχω λίγα σχόλια σχετικά με τους αριθμούς. Το απόλυτο επίπεδο είναι από τη μια μεριά και από την άλλη οι τάσει. Αυτό που εξηγήθηκε τώρα στην παρουσίαση ήταν οι τάσει για χώρες οι οποίες έκαναν πρόοδο, επέτυχαν πρόοδο σε πολύ μεγάλο επίπεδο, όπου βρισκόταν, βρίσκονταν όμως σε πρόβλημα πριν και άλλες οι οποίες είχαν ήδη υψηλό επίπεδο και βλέπουμε εκεί μια μικρή επιδείνωση, όπω η Σουηδία. Όμω, σε σύγκριση με το υπόλοιπο τη Ευρώπη, η Σουηδία πάντα βρίσκεται πολύ καλά με το 7%. Όπως είπε και η πρόεδρος, η Σουηδία είναι πρότυπο σε πολλά πράγματα. Στην παιδεία όμως όχι τόσο. Έχουν σημαντικά προβλήματα και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εξτάσεων πίζα. Και αυτό έχει σχέση και με την αποκέντρωση που έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και ανισότητες και μέσα στην ίδια την ε, Σουηδία, αν, ε, μέσα στις διάφορες κοινότητες δηλαδή, και ήδη κάνουν προσπάθεια να το αντιμετωπίσουν αυτό οι Σουηδοί. Σημαντικό επίσης είναι να τονιστούν τα διάφορα προβλήματα που έχουν σχέση με το μεταναστευτικό και για παράδειγμα με το παιδευτικό ιστορικό των γονιών δεν είναι δηλαδή ντε και καλά ότι είναι μετανάστε, αλλά έχει σχέση με το τι μόρφωση έχουν οι γονεί των παιδιών αυτών με μεταναστευτικό ιστορικό. Τώρα για τι τάσει των ε, διαφόρων χωρών. Αν εξετάσει κανεί τα θέματα αυτά και υπό τον φακό τη οικονομική κρίση, ε, οφείλει να πει ότι εμεί χαιρόμαστε για παράδειγμα που η Ισπανία έχει σημειώσει πρόοδο. Αυτό έχει σχέση και με το γεγονό ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το κίνητρο να εγκαταλείψουν τα αγόρια του σχολείου για να πάνε να εργαστούν στην οικοδομή, η οποία όμω στο μεταξύ βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία και πληρώνεται πολύ λιγότερο. Επίση, στην Ελλάδα πολλοί έμειναν στο σχολείο διότι για αυτού οικονομικά δεν είναι ελκυστική η αγορά εργασία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάνουμε μελέτε για να δούμε και τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Η Πορτογαλία για μα είναι παράδειγμα, το καλό παράδειγμα στην ε, ε, περίπτωση αυτή, διότι οι Πορτογάλοι έχουν προχωρήσει σε άσκηση πραγματικής ε, πολιτικής και στρατηγικής με πολύ στέρεα βάση και έχουν ε, ασχοληθεί και πολύ με τις λεπτομέρειες. Εμείς υποστηρίζουμε τις χώρες μέλη βεβαίως και χρηματοδοτικά. Πολύ σύντομα τώρα για τη χρηματοδότηση. Εκεί σε ό,τι αφορά τις δαπάνες παιδείας Είναι δύσκολο γιατί οι δαπάνες παιδείας κυρίως αφορούν τους μισθούς και αμοιβέ των διδασκόντων και αυτά δεν έχουν άμεση επιρροή στους δείκτες. Θα δούμε αν υπάρχουν μειώσεις των αποδοχών των διδασκόντων και αυτές οδήγησαν ενδεχομένως σε κάποιο αποτέλεσμα μείωσης ε, των, ε, μάλλον αύξηση του αριθμού των παιδιών που αποχωρούν από το σχολείο. Εν τέλει, υποστηρίζουμε, όπως είπα, και πριν και Ερασμοσύν και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την εγγύηση υπέρ των νέων. Και τέλος, το καλό νέο είναι, όπως είπε άλλωστε και η Πρόεδρος, σχετικά με τα έντυπα αιτήσεων. Έχουμε κάπως απλουστεύσει τα έντυπα αιτήσεων. Είχαμε και την ευκαιρία να το εξηγήσουμε αυτό. Μετά από την απλούστευση των διαδικασιών, έχουμε λάβει τώρα 40% παραπάνω αιτήσει και έχουμε μπορέσει να χρηματοδοτήσουμε 50% παραπάνω ε, τέτοια σχέδια. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος, πράγματι είναι θετικέ ειδήσει που μας ε, δώσατε. Δείχνει λοιπόν όντω ότι όταν απλουστεύονται οι διαδικασίες, κάθονται και οι άνθρωποι και γράφουν περισσότερες αιτήσει για χρηματοδότηση. Καλό αυτό. Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και θα πρέπει η Επιτροπή Πολιτισμού και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να ε, λάβει την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία έχετε στα σκαριά. Κυρία Βάντεν Χράφ, ευχαριστώ πολύ που περάσατε σήμερα από εδώ. Ε, σημειώστε, αυτό θα σας προτείναμε ούτως ή άλλως, να περιλάβετε στην τελική μορφή της μελέτης και το ερώτημα κατά πόσον τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεως έχουν συμβάλλει κάπως στη μείωση του αριθμού των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Να το σημειώσετε και αυτό λοιπόν. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τελική έκδοση της ε, μελέτης σας και ασφαλώς θα παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας, διότι το θέμα πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πολύ που μας εξηγήσατε τα προσωρινά πορίσματα της μελέτης σας. So, liebe Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε και άλλους ε, επισκέπτες, όπως βλέπετε εδώ, προσκεκλημένους. Οπότε, να σας παρουσιάσω τέσσερις νέους, οι οποίοι είναι η Διοικητική Επιτροπή ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να συνδέσει το θέμα της Ένωσης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα λέγεται Νέοι Ευρωπαίοι Δεσμευμένοι. Έχουμε εδώ την ε, Αμαντίν Λεβαγλέ που είναι η συντονίστρια. Τον Σιμό Μπουκερέλ είναι ο πρώτος ε, αρχισυντάκτης και η Λουσί Ζακλίν που είναι η αναπληρώτρια αρχισυντάκτης και ε, σας ευχαριστούμε καθώς και τον Τεό Γκουιτόν και σας ευχαριστούμε. Έχετε 15 λεπτά όπως ε, θέλετε. Μπορεί να κατανείμετε το χρόνο αυτό μεταξύ σα για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας και μετά έχουμε και ένα τέταρτο ε, συζήτησης. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. οποίο θέλει μπορεί να αρχίσει. Καλημέρα σας. Συγγνώμη, ε, ε, αισθάνομαι κάποια πίεση εδώ πέρα, δεν ξέρω τις ε, μεθόδους εργασία. θα χαλαρώσω όμω. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να συστηθούμε. Εγώ λέγομαι ο Τιό Γκουιτόν, είμαι 18 ετών, εργάζομαι στο επίπεδο των ενώσεων και συνεταιρισμών της νεολαίας και δημιούργησα τον πρώτο οργανισμό ε, και επίσης ασχολούμαι με το ε, ελεύθερο ραδιόφωνο στην περιοχή Σάρτε που είναι στην περιοχή του Λουάρ και κάνουμε προσπάθειες για την κατάρτιση των νέων και δηλαδή την κατάρτιση στη χρήση των νέων και είμαι αρμόδιος και για μια ένωση που λέγεται Diversity και προσπαθεί να βοηθήσει τους ε, νέους να ασχοληθούν περισσότερο με τα θέματα της Ευρώπης. Θα επανέλθω επ' αυτού. Καλημέρα σας. Λέγομαι Ρουσίου Ζακλίν, είμαι 17 ετών, είμαι ε, ε, μαθήτρια στο Λύκειο. Είμαι αρχιζεντάκτρια του πρόγραμματος αυτού και είμαι υπέρ της οικολογίας, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι η αρμόδια για την ε, Διεθνή Αμνηστία στο σχολείο μου και είμαι και επίσης αρμόδια για την εκπαίδευση σε μια εφημερίδα και ασχολούμαι και με τον ιστοχώρο La Ruche, η Κυψέλη. Λέγομαι Αμαντίν Λεβαρλέ, είμαι 18 ετών, είμαι τελειόφοιτη λυκείου όπως η Λουσί. Ασχολούμαι με ένα οπτικοακουστικό πρόγραμμα, δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Είμαι μέλος του Προεδρείου της ε, Ένωσης Γκέτρε που είναι μια ένωση για τους νέου τη υπαίθρου που ασχολείται με τα οπτικοακουστικά ασχολούμαι επίσης με διάφορα άλλα μέσα όπως την Κυψέλη το Λαρού που είναι για τους νέου και τους ε, ελεύθερου επαγγελματίε και επίσης με το Νοκταμπούλ. Λέγομαι Σιμών Μπουκρέλ, είμαι στη Λίλ στο Πανεπιστήμιο για πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Θα είμαι ο αρμόδιος για το ντοκιμαντέρ Συμμετέχω σε διάφορες ενώσεις, είμαι πρόεδρος της Κυψέλης αυτής και σε άλλα προγράμματα συμμετέχω και σε κάποιο συμβούλιο για την νεολαία. Alors, je vais vous présenter en quelques mots le projet. Λοιπόν, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Youth Europeans Involved. Φασιζόμαστε σε μια απλή διαπίστωση η νεολαία περιγράφεται ως ε, ιδιαίτερα ατομικίστρια και μακριά από την πολιτική και επίσης αναβλητική σε διάφορες χώρες. Όμως πρέπει να εκφράσει άποψη γιατί δεν υπάρχει εκτίμηση για τους νέους. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα ντοκιμαντέρ δύο ωρών για να δείχνει πόσο συμμετέχουν στη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νέοι για να συναντούμε με νέους παντού στην Ένωση οι οποίοι συμμετέχουν σε προσπάθειες για ανθρωπιστικές ε, αξίες και να δούμε πώς είναι το πλαίσιο του κόσμου των ενώσεων στην Ευρώπη. Ο στόχος μας είναι, πρώτα απ' όλα λοιπόν, θέλουμε οι νέοι να ασχοληθούν με την κοινή γνώμη, να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει αυτή τη συμμετοχή των νέων. Ο τίτλος μας είναι ακριβώς ε, κάτι που αντικατοπτρίζει αυτό, στηρίζει την προσπάθεια της Ένωσης ε, να ενταχθούν οι νέοι στην ε, δραστηριότητα, για τη δραστηριότητά της, της Ένωσης και να προτείνουμε λύσεις που να επιτρέψουν να ε, ενταχθούν ακόμη περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια. Τρεις ενώσεις ασχολούνται με το θέμα αυτό, όπου συμμετέχουν μόνο νέοι, που ε, ασχολούνται με θέματα δημοσιογραφίας και οπτικοακουστικά. Μέσω ενός τέτοιου προγράμματος θέλουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων στην Ένωση, στα κοινά και να δείξουμε και στην ευρύτερη κοινή γνώμη τι μπορούν να συμβάλλουν οι νέοι εάν είναι δυναμικοί και ασχολούνται με κοινοφελείς ε, στόχους. Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Να διευκρινίσουμε ότι δεν θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να περιοριστεί σε λίγους. Θέλουμε να βγει από τα γαλλικά σύνορα. Και αυτή την ευκαιρία θέλουμε από εσά, την ευκαιρία μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με όλες τις ενώσεις νέων στην Ευρώπη. Η Ένωση ε, Diversity που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα αυτό, εκεί όπου είμαι πρόεδρος από τότε που την δημιούργησα το 2017, έχει πολλά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τη μεγάλη εθνική συζήτηση της Γαλλίας. Η νεολαία να ξαναμπεί στο κέντρο αυτής της συζήτησης είναι η επιδίωξή μας και βλέπουμε ότι δεν συμμετέχουν αρκετά στον πολιτικό δημόσιο διάλογο οι νέοι. Ιδίω στην ε, μεγάλη αυτή συζήτηση που γίνεται τώρα. Ε, Στι 4 Μαρτίου, λόγω χάρη, θα οργανώσουμε μια εκδήλωση με νέου από οποιαδήποτε προέλευση στο ε, κοινωνικο-οικονομική, κάποιου που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, όπω και μαθητέ ε, του Λυκείου του Γυμνασίου ή κάποιου που ασχολούνται με τοπική πολιτική πέραν αυτών ε, έχουμε και άλλες επιδιώξεις. Κοιτάζουμε το τι θα γίνει με την ε, ιδιότητα του πολίτη στο σχολείο και την αγωγή του πολίτη και με το πόσο μπορεί να αποκτήσει πολιτική ταυτότητα νεολαία. Βλέπουμε σήμερα ότι οι νέοι ψηφίζουν λίγο. Δεν πάνε να ψηφίσουν αλλά δεν έχουν ε, ε, εκπαιδευτεί και γι' αυτό, δεν έχουν, δεν έχουν την απαραίτητη καλλιέργεια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε την πολιτική ταυτότητα των νέων στο σχολείο ήδη. Και μπορούμε να πάμε ακόμη παραπέρα. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα μπορούσε το δικαίωμα της ψήφου να δίδεται ήδη από τα 16 χρόνια της ηλικίας. Επιπλέον, έχουμε μια χάρτα, μια χάρτα συμβολικού χαρακτήρα που ζητούμε από του εκλεγμένου, ε, του τοπικού εκλεγμένου να την υπογράψουν, την χάρτα diversity, έτσι τη λέμε. Και έχουμε και άλλα προγράμματα, προγράμματα για όσου έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, σε συνεργασία με ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό σταθμό ενώσεων που προσπαθεί να οργανώσει ραδιοφωνικέ συνεντεύξει με όσου έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, οι οποίοι δεν έχουν άλλο τρόπο έκφρασή του. Και έχουμε και μια εταιρική σχέση ε, η οποία λέγεται Στούγεδα ε, που φέρνει σε επαφή δύο πόλεις, ε, τη μία στην Γαλλία κοντά στη Σάρτ και την άλλη στην Πολωνία. Στόχος είναι να δούμε και την στρατιωτική διάσταση τη νεότητα. Ε, σε συνδυασμό με τον πρόεδρο τη Πολωνία. Η ε, Κυψέλη δημιουργήθηκε το 2019. Είναι ένα διαδικτυακό μέσο επικοινωνία. Ε, συμμετέχουν νέοι 17-20 ετών από όλη την Γαλλία, από οποιαδήποτε κοινωνική και οικονομική προέλευση. Ένα ιστότοπο όπου δημοσιεύουμε συστηματικά άρθρα. Άρθρα που πρέπει όμω να σέβονται τη χάρτα των νέων δημοσιογράφων. Πρέπει να είναι ανθρωπιστέ και προοδευτικοί όσοι γράφουν και σύντομα ελπίζουμε να έχει και οπτικοακουστική κάλυψη ο ιστοτοπός μας με συζητήσεις, οργανωμένες συζητήσεις και ρεπορτάζ. Η τρίτη ένωση ε, ονομάζεται Getter Prod Get Prod στη ΣΑΡΤ στη Γαλλία. Ε, την διευθύνουν νέοι. Δημιουργήθηκε το 2016 από τον ΤΕΟ και σκοπός ήταν να δώσει οπτικοακουστικό υλικό σε όλους τους νέους, οποιασδήποτε προέλευσης, οποιοδήποτε κοινωνικού στρώματος και να αποκτήσουν μια έκφραση ως πολίτες από τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Πιλωτικής Διαχείρισης, την ε, Γενική Διεύθυνση την ε, έχει αναλάβει ο ΤΕΟ, ασχολείται με τις εταιρικές σχέσεις και τη χρηματοδότηση, καθώς και με την παρουσίαση του προγράμματος. Και ο ΤΕΟ δίνει τις γενικούς στόχους στις τέσσερις ομάδες της αρχής συνταξίας, ε, που είμαι εγώ υπεύθυνη, ασχολείται με τη σύνταξη των κειμένων και τη γραμμή που ακολουθεί η αρχή συνταξία, μετά τη διεύθυνση της Αμαντίν, που δεν είναι εδώ τώρα, που ασχολείται με την ε, καταγραφή και το μοντάρισμα των ε, φιλμ. Ο άλλος υπεύθυνο της Επιτροπής δεν βρίσκεται σήμερα εδώ και μετά υπάρχει και το θέμα της διοργάνωσης, τα διοργανωτικά, δηλαδή ποιος κάνει τι μέσα στο πρόγραμμα. Με αυτές τις συμπληρωματικές πληροφορίες θέλουμε να σας δείξουμε ότι είναι ένα πρόγραμμα νέων, από τους νέους για τους νέους. Ο στόχος της, πολιτικής, ε, της πιλωτικής επιτροπής είναι να συμμετέχουν νέοι από όλες τις όλα στρώματα, από όλες τις ηλικίε. Εγώ, ας πούμε, έχω αφήσει τη σχόλη μου για την ώρα και προσφέρω θελοντική εργασία στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι η νεολαία υπάρχει, είναι παντού και μπορεί να έχει παντού συμμετοχή για τα ντοκιμαντέρ και τα θέματα που θα αναπτύξουμε έχουν ένα βασικό αγώνα, ένα βασικό στόχο. Το θέμα της ισότητας, ιδίω μεταξύ των λαών, των κρατών μελών και των κοινωνικών κατηγοριών. Η πολιτιστική κληρονομιά της κάθε ευρωπαϊκής χώρας, η προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ιδιότητα του πολίτη, ιδίω των νέων, ο συσχετισμός με την ευρωπαϊκή θαγένεια, όπως έχει ονομαστεί ο όρος αυτός έχουν ε, τέτοιες προεκτάσεις στο πρόγραμμα Diversity. Και το βασικό είναι η συμμετοχή των νέων. Και βεβαίω εδώ αυτά απηχούνται και στη δική μα την Ένωση, το Λάριου. Επίση, ένα άλλο θέμα που θα αναπτυχθεί είναι η αλληλεγγύη και η ειρήνη. Σημαντικέ αξίε που θέλουμε να προωθήσουμε, καθώ και η οικολογία, η προστασία του περιβάλλοντο. Ένα θέμα που έχει τεράστια σημασία σήμερα, είναι επίκαιρο και έχει να κάνει και με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σε τέσσερις φάσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2019 για να βρούμε τη χρηματοδότηση και τις εταιρικέ σχέσεις, να γίνουν οι διάφορες περιβάσεις στα προγράμματα, η σύνταξη των κειμένων, η καταγραφή των φιλμ και το μοντάρισμα, μετά η οριστική παρουσίαση όσων έχουν γυριστεί, μετά Σεπτέμβριο με Ιούνιο 2020 του χρόνου, εκεί θα πάμε να γυρίσουμε στις διάφορες χώρες ουσιαστικά, επιτόπου. Τρίτη, Ιούλιος, Οκτώβριος 2020, δηλαδή εκεί θα γίνουν τα μοντάζ των ντοκιμαντέρια στη Γαλλία και θα αρχίσουν να προβάλλονται. Ε, τον Νοέμβριο του 2020 επιτέλου. Ελπίζουμε θα προβληθεί επισήμω σε πρεμιέρα και το ντοκιμαντέρ με τη Συμφωνία των Λοιπόν, ο προπολογισμό. Τον προπολογισμό τον έχει υπολογίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Και όλε οι επιτροπέ συμμετείχαν. Έχουμε προβλέψει τα εξή. 1500 ευρώ. 35 μάλλον χιλιάδες ευρώ για τα οπτικοακουστικά, που είναι δυστυχώς πάντοτε ακριβά, και είναι δύσκολο οι νέοι να γυρίσουν ταινίε ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Η επικοινωνία 7.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι η επικοινωνιακή πολιτική δεν είναι αμεληταία. Και η διοργάνωση. Τα ταξίδια, οι ομάδε που θα αναλάβουν το γύρισμα. 82.500 ευρώ είναι ο προηγούμενο μα προπολογισμό. Και σε σύγκριση με τα επαγγελματικά ντοκιματέρ που γυρίζονται, α πούμε, είναι πολύ χαμηλότερο ο προπολογισμό μα. Ήταν και επιλογή μα αυτό. Θέλαμε να εξοδέψουμε λιγότερα, διότι θεωρούσαμε ότι δεν έχουμε και τι δυνατότητε να εξοδέψουμε παραπάνω. Ναι, να συμπληρώσω. Συνεργασία με του ευρωπαϊκού θεσμού. Το πρόγραμμα European Youth Involved είναι βαθιά ευρωπαϊκό και βαθιά ριζωμένο στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Με την βούληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει την νεότητα στο κέντρο των πολιτικών τη στην καρδιά της χάραξης πολιτικών. Χρειάζεται συνεργασία και στο επίπεδο το οικονομικό όμως. Σε ένα επίπεδο διοργάνωσης και θεσμικό. Εμείς δεν είμαστε καθόλου κατά της Ευρώπης και με συγχωρείτε κιόλα για την έκφραση. Είμαστε βαθιά Ευρωπαίοι και φιλοευρωπαϊστές. Οπότε για μάς είναι προτεραιότητα να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διότι θεωρούμε ότι μπορούμε να παραμείνουμε ουδέτεροι, συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να είναι υπέρ των όσων προτείνουμε, είναι υπέρ των νέων. Ε, μιλάμε για ενώσει νέων, αλλά για να γράψει κανεί ένα άρθρο σε μια εφημερίδα ή απλώ να εκφραστεί ή να έχει βήμα για να εκφραστεί, είναι δύσκολο. Πρέπει να έχει κάπου μια επίσημη συμμετοχή. Γι' αυτό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν γίνονται σχόλια, πολλές φορές λέμε ότι αποτελεί μία ανάληψη ευθύνη, δηλαδή να εκφραστεί κανείς επισήμως και υπέρ της Ευρώπης και των νέων που έχουν πολλά να πούν και θέλουν να εκφραστούν για πράγματα που τους είναι σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακή παρουσίαση. Μα εσείς οργανωμένοι σαν ένας ε, μικρός ε, ραδιοφωνικός σταθμός με πολύ επαγγελματικό τρόπο πολύ ε, αξιέπαινο πολύ επαγγελματικό πολύ δέσμευση οπότε αυτές οι, αυτές οι φήμες που ακούμε ότι οι νέοι είναι απολύτικοι ότι δεν συμμετέχουν στα κοινά δεν ισχύει Αντίθετα, είστε ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι και ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι για τα κοινά. Το εγχείρημά σας το δείχνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι. Πρώτη η Σίλβια Κώστα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πραγματικά μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Υπέροχο πρόγραμμα υπέροχο σχέδιο με πολύ σαφείς στόχους, φανταστικά διαρθρωμένο σε όλη του την ε, περιγραφή. Μας είπατε τα χαρακτηριστικά. Ε, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε μια ταυτότητα ευρωπαϊκή κοντά στους νέους της γενιάς σας και όχι σε αντιδιαστολή με τις άλλες γενιές. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των νέων, της εθελοντικής εργασίας, της ευρωπαϊκής ε, νεολαίας που θα έχει ε, ενεργό συμμετοχή στα πράγματα, τα πολιτικά πράγματα, είναι σημαντικό. Γι' αυτό θα το σήμερα, γιατί κλείναμε και το Erasmus Συν και την Δημοτική Ευρώπη. Όλα αυτά είναι σχετικά. Είναι δυνατότητες για σας στο μέλλον να συμμετέχετε, διότι υπάρχουν πολλές αναφορές στα προγράμματα αυτά που θα ξεκινήσουν το 2021, Μερικά έχουν ήδη ξεκινήσει βεβαίως, ε, λειτουργούν, αλλά αυτό για τα οπτικοακουστικά, η πρόθεση της ε, ενεργού πολιτικής μετοχή αυτό της Δημιουργικής Ευρώπης και εκεί έχουμε προβλέψει στήριξη της δημοσιογραφίας και των νέων. Ή στα δίκτυα, τα ραδιοφωνικά και τα ε, άλλα μέσα, υπό την ευρεία έννοια τους, που είναι ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Θυμίζω επίσης το είπαμε, ε, έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς και δύο νέοι στο Στρασβουργό, οι οποίοι ήταν τη δικτύου γιουροφόνικα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε εταιρικέ σχέσεις. Ένα παράδειγμα στη χώρα μου υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία φιλευρωπαϊστών νέων, η Ουτοπία, ένα online περιοδικό, ε, θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή για να γνωριστείτε κιόλα. Εσεί διαλέγετε για να δείτε τι γίνεται σε αυτό το χώρο, γιατί δεν είναι και πολλοί μήνε για να κλείσουν οι συνεργασίε. Και θα κλείσω με αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε κι εσεί οι ίδιοι ότι θέλετε να δουλέψετε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε. Η εκστρατεία που έκανε το Κοινοβούλιο για την ευαισθητοποίηση των νέων ε, Σα άγγιξε και εσείς τι συμβουλές θα είχατε να δώσετε όχι για να γίνει εκστρατεία προκλοκή των κομμάτων και των πολιτικών ομάδων αλλά για να ε, ευαισθητοποιηθούν οι νέοι ως προς την ενεργό άσκηση της πολιτικής τους ιδιότητας. Έχετε απάντηση. Ε, τη ερώτηση. Είμαι νέο. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Το ιδανικό θα ήταν να συμμετέχουν όλοι οι νέοι. Ποιο θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο αντίκτυπο, ε, στην περιέργεια, τη φιλομάθεια, τη διάθεσή σα για μάθηση σε σχέση με το κάνουμε και. Ε, υπάρχει προσδοκία για ευρωπαϊκό περιεχόμενο για εσά από ό,τι φαίνεται στα προγράμματά σας. Κοιτάξτε, κάποιες φορές τα πράγματα αυτά είναι λίγο θολά για μερικούς νέους. Θα πρέπει να συνδυάσουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Μερικές φορές τα πράγματα είναι πολύ θεσμικά και πολύ θολά. Εγώ έρχομαι από περιοχή της Πέθρου. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ είναι λίγο απρόβλεπτο, μη αναμενόμενο. Μιλάμε για νέους που δεν είναι απλώ ότι δεν ενδιαφέρονται, μπορεί να μην ενδιαφέρονται με το σωστό τρόπο. Έχει αλλάξει η προσέγγιση. Οι νέοι θέλουν κάτι που να του αγγίζει απευθεία. Θέλουν να συμμετέχουν. Απλώς οι προσεγγίσει κάποιες φορές είναι πολύ περίπλοκε ή πολύ αφηρημένες. Ευχαριστούμε, Ζαμπίνε Φερχάιερ. Και εγώ με ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας. Αυτή την ε, προσπάθεια αφιλοκερδός ε, να συμβάλετε. Δεν είστε επαγγελματίε, αλλά ε, εργάζεστε με επαγγελματικό τρόπο. Βεβαίως δεν ασχολείστε μόνο με το να καλέσετε τον κόσμο να ψηφίσει, αλλά να συμμετάσχει ευρύτερα. Λέτε ότι θέλετε η προπαρασκευαστική φάση να είναι μέχρι τον Αύγουστο και να λήξει τον ε, Νοέμβριο του 20. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με τι εκλογέ. Να δείξετε στου νέου, θέλετε, τι δυνατότητε υπάρχουν για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια του ευρωπαϊκού εγχειρήματο στην Ευρώπη. Ερώτηση. Θα πάτε σε διάφορε χώρε. για να δείξετε πώ συμμετέχουν οι νέοι με διαφορετικό τρόπο εγώ στη δουλειά που κάνω με τους νέους, στα σχολεία και σε άλλα πλαίσια, είναι ότι πολλοί νέοι δεν ξέρουν πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν, πού θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Θα μπορούσατε λοιπόν να βοηθήσετε, να τους δώσετε στοιχεία στους νέους, να δούνε τι μπορούν να κάνουν, τι υπάρχει γύρω τους, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Λέτε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με την Κομισιόν να συνεργαστείτε με εθνικές οργανώσεις νέων, με διάφορες ε, ενώσεις νέων γενικότερα. Αυτό θέλετε ή κυρίως θέλετε να συνεργαστείτε κατά, καταρχάς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι και σε εθνικό επίπεδο μπορείτε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Όντως, οι νέοι δεν έχουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν, δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν, πώ να συμμετάσχουν. Έτσι διαπιστώσαμε και εμεί ότι έχει κατάσταση. Όλοι μόλι ε, τελειώσαμε το Λύκειο ή είμαστε ακόμη στο Λύκειο. Κανεί δεν μας μαθαίνει πώ να βοηθήσουμε, πώ να συμμετάσχουμε. Να σα πω κάτι προσωπικό. Πήγα σε ένα μικρό λύκειο στην Ήπεθρο με 300 ε, μαθητές και παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να κάνω πολλές απουσίες πήρα το απολυτήριό μου, το μπακ με καλό βαθμό Παρά το ότι δεν ε, εντάχθηκα πλήρω ε, στην ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως την προβλέπει το σχολείο. Πρέπει οι νέοι να μάθουν πώς να συμμετάσχουν, να δημιουργήσει κάτι μια ένωση, να συμμετάσχει σε ένα εγχείρημα, να χτυπάει πόρτες. Είναι δύσκολο για ένα νέο. Τι δυνατότητες υπάρχουν λοιπόν οι νέοι να συνεργαστούν. Συμμετέχουμε στο Εθνικό Δίκτυο του Τύπου για την Νεολαία. αφού έχει ένα ευρύτερο δίκτυο. Δεν νομίζουμε τόσο δύσκολο να κινητοποιήσουμε τους νέους. Έχουμε ήδη 40 που εργάζονται εθελοντικά και αφιλοκερδός για μας, πέρα από τα μέλη της δικού σας επιτροπής. Και φυσικά θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία. Δεν θέλουμε να ασχολούμεθα μόνο με τους νέους. Ούτε να λέμε ότι οι νέοι είναι οι καλύτεροι. Λέμε απλώς ότι οι νέοι έχουν και αυτοί το ρόλο τους. Αλλά και οι μεγαλύτεροι έχουν την πείρα τους, μπορούν και εκείνοι να βοηθήσουν. Αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουν τους νέους. Αυτό που λέγεται ότι είμαστε οι πολίτες ε, του αύριο, αυτό είναι αλήθεια. Ε, η πρόεδρο σας ευχαριστώ. Η Julie Ward. Τι ωραία που είστε εδώ. Σας άκουσα να μιλείτε για την ειρήνη. Είπατε ότι δουλεύετε υπέρ της ειρήνης και διερωτώ με αν γνωρίζετε ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011 υπογράφτηκε μια δέσμευση για την ειρήνη. Ούτε πολλοί ευρωβουλευτές δεν το ξέρουν αυτό. Και θα σας παροτρύνω να το διερευνήσετε και να προσπαθήσετε να το καταστήσετε γνωστό και σε περισσότερους ανθρώπους αυτό το Peace Project. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έλαβε το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης το 2012 και ε, αυτό που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το γνωρίσουν και όλοι οι ευρωβουλευτές που θα έρθουν εδώ να καταλάβουν τις ε, έδρες. Και αυτό έχει και κάποια σημασία για τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής προσπάθειας. Έχω και άλλες πληροφορίες για λογαριασμό σας. Υπάρχει μια θαυμάσια ε, οργάνωση που λέγεται International Children Press Center ε, που ασχολείται με παιδιά μέχρι ε, την ηλικία του εφήβου και τους δίνει βάσεις για να μπορέσουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Αυτοί έχουν έδρα στο Άμστερνταμ τη Ολλανδία και ασχολούνται πολύ και εδώ στο Κοινοβούλιο και θα χαρούν πολύ να έχουν επαφή μαζί σα οι άνθρωποι αυτοί συμμετέχουν σε ένα πολύ ενδιαφέρον project στο Άρανταλ της Νορβηγίας. Είναι μια θαυμάσια εβδομάδα που όλοι εκεί συνέρχονται και μιλούν για πολιτική, για ε, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την πολιτική και τους πολιτικούς. Νομίζω ότι και αυτό θα σας ενδιαφέρει. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ επιθυμεί κανεί εκ των ε, νέων. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρότασή σα Είμαι βέβαιο ότι θα μας ε, βοηθήσει πάρα πολύ. Επανέρχομαι στο θέμα της Ειρηνή. και αυτό που έχει ενδιαφέρον να μιλεί κανεί για ειρήνη, μιλούμε συχνά για διεθνή ειρήνη. Όμως η ειρήνη παίζει ρόλο και στο τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, κατά τη παρενόχληση στο σχολείο, κατά για τον αγώνα γενικότερα κατά των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων που αισθάνονται μόνοι τους, που είναι διαφορετικοί. Και η ένωση μας λέγεται diversity, δηλαδή ε, πολυφωνία, ας ε, πολυφωνία πολιτισμική για παράδειγμα. Και αυτό παίζει ρόλο και νομίζουμε ότι η ειρήνη και πέρα από αυτό, μιλούμε για διεθνή ειρήνη βέβαια, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για αυτή την ειρήνη στο σχολείο, στο μικρό χωριό, όπου διαμορφώνονται πολλές καταστάσεις. Δίνω και μια προσωπική νότα. Ο δήμαρχος της κοινότητάς μου με αντιπαθεί. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Και εδώ και τρία χρόνια με κατηγορεί για ε, ε, δίθεν παράνομα πράγματα κλπ. Και έχω ναι. ζητήσει κατ' να το δω και ποτέ δεν με δέχθηκε. Είναι και αυτό ένα είδο ειρήνη, ωστόσο, πρέπει να αποκατασταθεί. Ορίστε, σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε, για την σημαντική αυτή υπόδειξη ότι η ειρήνη ξεκινά και από ε, εμάς τους ίδιους ε, στο προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ακούσατε και πολλές χρήσιμες συμβουλές από τους συναδέλφους μου για το τι μπορείτε ακόμη να κάνετε, ποιες συνεργασίες να επιδιώξετε. Χαίρομαι που έχουμε κοντά μας και τον κύριο Αμπαμόντε που είναι αρμόδιος για το Creative Europe Program και για το ε, τμήμα εκείνο που αναφέρεται στην εργασία των media και είμαι βέβαια ότι ε, θα υπάρξει ίσως και κάποια δυνατότητα χρηματοδότησης για το σχέδιο που ε, προωθείτε εσείς, το project σας δηλαδή. Και το Media Desk στη Γαλλία είναι βέβαια ο πρώτος σας που μπορεί να σας βοηθήσει, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον που και ο κύριος Σαλβαμόντε παρακολούθησε την παρουσίασή σας εδώ, της Επιτροπής δηλαδή. Και ίσως και ίσως ε, μπορείτε να διασφαλίσετε και κάποια υποστήριξη ας πούμε και από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Άρτε και όταν το φιλμ σας θα είναι έτοιμο μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, και εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε ενδεχομένως στην αποκατάσταση σχέσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, εξηγήσατε και παρουσιάσατε το project σας. Νομίζω ότι ακούσατε και από εμάς πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το project αυτό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και Εάν χρειάζεστε κάποια χείρα βοηθείας, πολύ ευχαριστώ να ε, σας δεχθούμε, εάν το θεωρείτε ε, αναγκαίο. Και όπως είπα και πάλι, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστίες από τους τέσσερις νέους. Wir Αμέσως συνεχίζουμε, λέει η Πέτρα Κάμερ Εβερτ. Επιτρέψτε μου μια στιγμή να ε, αποχωρήσω και θα επανέλθω αμέσως γιατί δεν αντέχω. Αγαπητέ και αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τώρα με την ε, συνεδρίασή μας. Μας μένει περίπου μισή ώρα. Έχουμε το επόμενο θέμα τη ημερησίας διατάξεως μα που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση των μέσων ενημέρωση στην Ουγγαρία που ω γνωρίζετε προεβδομάδο, ιδρύθηκε ε, ίδρυμα, κέντρο ευρωπαϊκό ίδρυμα, ε, ich ε, nicht nur diese και είναι κάπως ανησυχητική κατάσταση γιατί έχει και δραματικές επιπτώσεις στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και επομένως και στα θεμέλια της δημοκρατίας. βιώνουμε πράγματι τώρα μια νέα κλιμάκωση των σχέσεων Τη επιδείνωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουγγαρία και θα έχετε ακούσει και τις δηλώσει του Πρόεδρου της Επιτροπής ε, ε, Jean-Claude Juncker και νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε πράγματι μια δύσκολη κατάσταση είχαμε έχουμε άλλωστε ήδη ψηφίσει σχετικό ψήφισμα και είχαμε ζητήσει τότε την την, ε, ε, την ε, επιβολή των διατάξεων του άρθρου 7 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των μέσων ενημέρωσης στην χώρα αυτή, στην Ουγγαρία. Όπως είπα, θεωρούμε την κατάσταση ενισχυτική, την παρακολουθούμε προσεκτικά βεβαίω ε, εξαρτώμεθα από ε, τα διαφορά άρθρα στι εφημερίδε για την ενημέρωση. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θετικό το ότι βρίσκεται κοντά μα ο κύριο Σάμπα Μόντε σήμερα και θα μπορέσει να μα εξηγήσει και να ακούσουμε δηλαδή από τα χείλη του τα ε, σχετικά και το ποια δράση προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία του ευρωπαϊκού δικαίου στην χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Σας καλωσορίζω όλους. Προσπαθήσαμε να έχουμε κάποια στοιχεία για τη δημιουργία αυτού του ομίλου μέσων. Τέλη Νοεμβρίου λοιπόν πέρυσι, πάνω από 12 διοκτήτες μέσων μετέφεραν 470 ε, περίπου μέσα σε αυτό το κέσμα. Όλα τα μέσα αυτά ήταν ιδιωτικά. Όλα αυτά τα μέσα συμπεριλέμβαναν ε, website ειδήσεων, εφημερίδες, κανάλια τηλεόρασης, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ε, ταμπλόιντ εφημερίδες, εφημερίδες, αθλητικές εφημερίδες, διάφορα περιοδικά και όλες τις περιφερειακές εφημερίδες της χώρας είναι σημαντικό ότι αυτό το κέσμα, αυτό το ίδρυμα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κανονικός ε, οργανισμός, ίδρυμα δηλαδή, με βάση τον ε, Ουγγρικό Αστικό Κώδικα και ελέγχεται από την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι έχουν ε, σχέση με το ΦΙΝΤΕΣ, το κυβερνητικό κόμμα. Μέσω ενός διατάγματος ο ρυθμιστικός οργανισμός, το Συμβούλιο για τα Μέσα και η Αρχή Ανταγωνισμού αποκλείστηκαν από την εξέταση αυτής της συγχώνευσης ε, λόγω του ότι αυτή η διαδικασία έχει στρατηγική εθνική σημασία. Προσπαθήσαμε να δούμε τι επίπτωση είχε αυτή η διαδικασία στο τοπίο των μέσων στην Ουγγαρία και αφετηρία της ε, αξιολόγησής μας είναι ένα ανεξάρτητο μέσο που λέγεται επιθεώρηση των μέσων που γίνεται από το Ινστιτούτο της για την ε, πολυφωνία των μέσων που καθορίζει κριτήρια για την πολυφωνία των μέσων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη. Είχαμε μια έκθεση για την Ουγγαρία το 2017. Ήδη έκθεση αυτή πριν από τη δημιουργία του ΚΕΣΜΑ λοιπόν αυτού Αναφέρονταν διάφοροι κίνδυνοι που το μέσου ή ε, πολύ ψηλού επίπεδου για τον πλουραλισμό των μέσων. Ιδιαίτερα. Η συγκέντρωση ιδιοκτησία μέσων ήταν υψηλό κίνδυνο, 70%. Είχε δηλαδή εκτίμηση υψηλού κινδύνου, βαθμολόγηση. Λόγω διαφορετικών αδυναμιών ε, του νόμου και της έλλειψης ενός ε, γνησίως ανεξάρτητου ρυθμιστικού οργάνου, ρυθμιστικής αρχής. Αυτά τα έλεγε ήδη η επιθεώρηση μέσων. Και όσον αφορά τη συγκέντρωση ε, μέσων διαφόρων ειδών, η ίδια μελέτη έλεγε ότι λόγω της ε, σημερινής πολιτικής κουλτούρας τα περισσότερα μέσα παράγουν το ίδιο περιεχόμενο που είναι φιλικό προς την κυβέρνηση. Λόγω αυτής της νέας διαδικασίας ο κίνδυνος αυτός θα γίνει ακόμη σοβαρότερος. η επιρροή των ιδιοκτητών ή ε, της οικονομίας επί του περιεχομένου των μέσων θεωρείται επίση υψηλή 67%. Η πολιτική ανεξαρτησία των μέσων ε, θεωρεί το μέσο επίπεδο 63%. Διότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πολιτική και τα πολιτικά κόμματα ασκούν άμεση ή έμεση επιρροή και έλεγχο επί των μέσων. Και τέλος, ο υψηλότερος κίνδυνος, ο πολύ έντονος κίνδυνος, 97% βαθμολόγηση, είχε να κάνει με το ρόλο του κράτους για την χρηματοδότηση και τον έλεγχο των μέσων. Κατά πάσα πιθανότητα η δημιουργία αυτού του Ιδρύματος Κέσμα θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το τοπίο των μέσων στην Ουγγαρία. Μια μεγάλη ανησυχία είναι πώς θα γίνονται οι κρατικές ανακοινώσεις και διαφημίσεις μέσω του τύπου κατά πάσα πιθανότητα θα δίδεται σε φιλοκυβερνητικά μέσα και όχι σε επικριτικά μέσα. Και θα αυξηθεί λόγω αυτής της διαδικασίας ε, η συγκέντρωση αυτών των ε, χρηματοδοτήσεων. Άρα τα ανεξάρτητα μέσα θα έχουν ε, ακόμη λιγότερη πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση, άρα περαιτέρω στρέβλωση της αγοράς. Στην απάντηση που σας στείλαμε μετά την ερώτησή σας, ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς ανέφερε το θέμα ότι έχει θυγεί το θέμα αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας ε, κράτους δικαίου. Έγινε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 11 και χθες. Ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς είπε ότι η δημιουργία του ΚΕΣΜΑ είναι άλλη μια ανησυχητική εξέλιξη. Τα θέματα των μέσων λοιπόν είναι υψηλή προτεραιότητα στη διαδικασία του άρθρου 7. Και είναι στο κέντρο της συζήτησης. Χθες όλα τα κράτη-μέλη που παρενέβησαν συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασαν ανησυχία για αυτή την εξέλιξη. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη, το γνωρίζετε ήταν στην απάντηση, ο, να συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέταση και τα θέματα. Τι έκανα. Ζήτησα από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας να δει αυτή τη διαδικασία και τι επίπτωση έχει στο τοπίο των μέσων και να κάνει μία μελέτη αντικτύπου με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσής της του 17. Βεβαίως είναι διατεθειμένοι να το κάνουν και θα το κάνουν τις επόμενες μέρες, τάχιστα. Και τα αποτελέσματα της μελέτης φυσικά θα τα λάβετε. Θα εξετάσουμε την κατάσταση και με βάση το άρθρο 30, παράγραφοι 1 και 2 τι νέε οδηγίε για τα οπτικοακουστικά μέσα που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ για τα οπτικοακουστικά πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από τι κυβερνήσει του και να, και να ασκούν τα καθήκοντά του με βάση του στόχου τη οδηγία. Ιδιαίτερα προωθώντας την ε, πολυφωνία των μέσων και τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος για την παρουσίασή σας που δεν μας χαροποιεί φυσικά. Καλό είναι που το Ινστιτούτο της Φλόρεντίας κλήθηκε να κάνει μία νέα μελέτη. Η ερώτησή μου. Θεωρείτε ότι από πλευρά ε, νομοθεσίας για τα καρτέλ, δηλαδή νομοθεσία ανταγωνισμού, υπάρχει δυνατότητα να παρέμβουμε γιατί το δίκαιο του για τα μέσα είναι περιορισμένο. Δεν υπάρχει νόμος για την συγκέντρωση των οπτικοακουστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ο νόμος για τον ανταγωνισμό. Ξέρουμε ότι η Ουγγαρία άλλαξε την νομοθεσία της όσον αφορούσε τη διαφήμιση. Αυτό βεβαίως αφορούσε ένα ιδιωτικό μέσο όπου μπορέσαμε να παρέμβουμε μόνο με το δίκαιο του ανταγωνισμού και την υποχρεώσαμε την Ουγγαρία να αλλάξει την ομοθεσία της. Βλέπετε μήπως μέσω αυτής της δυνατότητας να έχουμε κάποιες δυνατότητες. Μήπως θέλετε να απαντήσετε καταρχάς αυτό και μετά να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Βεβαίω, είμαστε σε επαφή με τους Ούγγρους συναδέλφους σε όλες τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις και η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε, τουλάχιστον από τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ, είναι βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών να πούμε ότι βάσει των κανονισμών περί συγχωνεύσεων η δημιουργία του ΚΕΣΜΑ δεν ε, μπορεί να ε, είναι κάτι που θα το εξετάσουμε εμείς. Η δικαιοδοσία της συναλλαγής είναι θέμα των εθνικών αρχών της Ουγγαρίας. και διέπεται από του εθνικού του κανόνε. Ο κανόνα για τα καρτέλ τη συγχωνεύση δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να ελέγξει ε, την απόφαση των Ουγγρικών αρχών να εξαιρέσουν αυτή τη συναλλαγή από την εφαρμογή των κανόνων για των κανόνων για τις συγχωνεύσεις, κατά των συγχωνεύσεων. Η συμπεριφορά ή οι πρακτικές του Ιδρύματος αυτού μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο των κρατών μελών, βέβαια, οπότε τότε θα ε, περάσουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ανταγωνισμό. Τότε και η Ουγγαρία και όπω τα άλλα θα πρέπει να σεβαστεί του κανόνε ανταγωνισμού, ιδίω ε, για τον έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων ή βοηθειών. Νομίζω ότι απαντήθηκε η ερώτησή μου. Είχε να κάνει με το θέμα τη πολιτική ανταγωνισμού, το δίκαιο ανταγωνισμού. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, που έχουμε του ομίλου Bertelsmann και Springer, αλλά όλα αυτά δεν είναι υποκρατικό έλεγχο. Άρα στην πραγματική ερώτηση. Ο κρατικός έλεγχος που υπάρχει αυτού του Ιδρύματος σε τι βαθμό επηρεάζει τη δουλειά των δημοσιογράφων. Έχουμε κάποια στοιχεία από αυτού. Πώς, πώς εκφράζεται συγκεκριμένα ο έλεγχος αυτού του Ιδρύματος. Ο κύριος Αμπραμόντε Ο έλεγχος εικάζεται ότι δεν είναι σαφής. Όλα τα, κράτη του, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν σχέση με το κυβερνοκόμμα. Διαπλοκή. Τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρω να σας πω. Ένας αριθμός ανθρώπων έχουν διασυνδέσεις με τον Ορμπάν και ήταν και δωρητές. Έφεραν αυτά τα μέσα, τα οπτικοακουστικά, στο Ίδρυμα. Είναι οικειοθελής δωρεά από την πλευρά των δωρητών των ε, συμμετεχόντων στο Συμβούλιο. και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πρώην βουλευτέ ή άλλοι που έχουν ε, διαπλοκή με την ε, κυβέρνηση. Για τον έλεγχο λοιπόν της κυβέρνησης επί το Ιδρύματος, μάλλον είναι σημαντικός, αλλά υποκρυπτόμενος. αλλά άρα δεν υπάρχει άμεσος κυβερνητικός έλεγχος για τα άτομα που είναι μέλη του ίδιου κόμματος. Ευχαριστούμε Σίλβια Κώστα. Ε, νομίζω η απάντηση πάντοτε είναι πιο δυσάρεστη στην Ουγγαρία. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Υπάρχει κλιμάκωση στο θέμα των μέσων. Να θυμίσω γρήγορα το 2017 ο νόμος για τις διαφημίσεις και τους φόρους 5,553. Μεγάλη πίεση στα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρώτο σημείο. Δεύτερο, η κρατική τηλεόραση ε, απέστειλε μηνύματα ε, της κυβέρνησης κατά και των προσφύγων. Έπειτα έκλεισε η πιο σημαντική δημοσιογραφική έδρα στην Ουγγαρία και τέταρτο, ακόμη και αν ήταν ελεύθερη συμμετοχή, υπήρχε εκβιασμός όπως λέμε στην ε, Ιταλία. Δηλαδή η διαφημιστική βάση περιορίστηκε και όλοι αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν, άρα κλείσανε πολύ. Αυτό από πολιτικής άποψη συνέβη ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο που την ε, στήριξε είχε ξεκινήσει, η διαδικασία του άρθρου 6. Είναι σοβαρά τα πράγματα από πολιτικής άποψη. Υπάρχει διαφορία ως προ το σημείο αυτό όμως. Και πρέπει να πω και το εξή σε σχέση με τους νόμου για την παρακολούθηση που έγινε από, το, από τη Φλωρεντία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν είναι ανεξάρτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί μπορεί να παρέμβει. Έχει δικαίωμα παρέμβασης να πει ότι η ανεξαρτησία απαιτείται για τις αρχές. Γιατί, γιατί αλλιώς είναι στον έλεγχο της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε κυρία Μπραμόντε. Θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε μόλις εφαρμοστεί η οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Για πρώτη φορά η οδηγία αυτή προβλέπει απέτηση ρυθμιστική ανεξαρτησία ανεξαρτησίας ενό το τόπου, ανεξαρτησία και στη λειτουργία του. Η οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά πρέπει και να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Στα τέλη του 2020 θα δούμε τι θα γίνεται. Τότε θα αρχίσουμε να το ψάχνουμε το θέμα. Τώρα δεν μπορούμε. Ιδίω στην περίπτωση του έργα. Ναι. Ευχαριστούμε. Έχω και άλλου συναδέλφου που θέλουν το λόγο. Αλλά πρέπει να κοιτάμε και το ρολόι. Ένα λεπτό καθένα αν γίνεται. Η ε, κυρία Σαρχεντίνη. Που ήταν ησυχήτρια στην αρμόδια επιτροπή γιατί η κατάσταση στην Ουγγαρία είναι τώρα κοντά μα, Αν συμφωνείτε, διότι βέβαια ε, μέλη εταίρων επιτροπών κατ' εξαίρεση λαμβάνουν το λόγο. Πάντω, πολύ ευχαριστώ αν συμφωνούν και οι υπόλοιπε ε, συνάδελφοι. Πρώτα ο κύριο Σβέρ. Για ένα λεπτό σα παρακαλώ κύριε. Ευχαριστώ αγαπητή πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο ε, για να θέσω μια ερώτηση. Πρώτα, οφείλω να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος που η δική μας Επιτροπή επικρίνει μια χώρα, μάλλον μια κυβέρνηση χώρας μέλους. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ποια κυβέρνηση θα επικρίνεται. Σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς, στην ε, Ουγγαρία η κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πιο ισορροπημένη από ό,τι στη Σλοβενία. η εκπροσώπηση δηλαδή πολιτικών απόψεων είναι πιο ισορροπημένη. Με ποιο τρόπο λοιπόν επιλέγετε ποιες κυβερνήσεις θα επικρίνετε. Μου φαίνεται ότι η ερώτησή σας απευθύνεται μάλλον σε εσάς. Σε, μάλλον σε μένα, με συγχωρείτε. Α, όχι, στον κύριο Αμπαμόντε, ωραία. Εσείς κύριε Αμπαμόντε, με ποια κριτήρια επιλέγει η ε, Κομισιόν Κυβερνήσει τις οποίες επικρίνει. Κοιτάξτε, έχουμε το Media Monitor Έχουμε Media Pluralism Monitor. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο καλύπτει, ένα μηχανισμό αν θέλετε, που καλύπτει όλες τις χώρες μέλη. Και κάτι, ας πούμε, είναι μια ανάλυση, μια συγκριτική ανάλυση οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων σε διάφορες χώρες μέλη. Αυτό που προκύπτει από αυτό το monitor είναι ότι καμιά χώρα μέλος δεν είναι απολύτως ε, οχυρωμένη απέναντι στους κινδύνους η κατάσταση το 2017 στην Ουγγαρία, όπως είπα προηγουμένως, ήταν ας πούμε πιο επικίνδυνη από την άποψη αυτή και ιδίω ε, η κρατική νομοθεσία περί χρηματοδοτικών ενισχύσεων στον τομέα των media Δηλαδή ε, μια ετεροβαρής ας πούμε ε, η μονομερής κατά κάποιο τρόπο στήριξη κάποιων ε, μέσων ενημέρωσης και πολύ, σε πολύ ψηλό. Υπήρχαν και άλλοι ε, παραμετροί όπως η συγκέντρωση ε, στα χέρια λίγων εμπορικές ή άλλες επιρροές, πολιτική εξάρτηση των μίδια. Λοιπόν, λαμβάνονται υπόψη πλήωνα κριτήρια και λόγω των εξελίξεων αυτών ζητούμε από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας να βασιστεί στην ανάλυση που έχουμε κάνει το 2017 για να εξετάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση σε ομίλους βελτιώνουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πολυφωνία των μέσων ή την επιδεινώνουν. Στην Ουγγαρία πάντοτε. Και οι κίνδυνοι αυτοί πρόκειται να ε, χειροτερεύσουν ή μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί. Ευχαριστώ Πολύ, λέει η Πέτρα Κάμερ Εύερτ. Υποθέτω ότι ω θεματοφύλακα των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλε τι χώρε μέλη εάν τηρούν τα προβλεπόμενα από τι συνθήκε και ενδεχομένω αναλαμβάνει και δράση ανεξαρτήτως του περί ποιας χώρας πρόκειται. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ, υπάρχουν χώρες μέλη ωστόσο όπου τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι παρημείνει, δηλαδή στην Ουγγαρία, όπως για παράδειγμα στην Σοβακία ή στη Μάλτα, όπου σημειώθηκαν και φόνοι δημοσιογράφων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφορες, διάφοροι όμιλοι, διάφορα, διάφορες εταιρείε χαρτοφυλακίων όπου περιλαμβάνουν και μέσα ενημέρωσης. Μπορώ να αναφέρω ακόμη και τον Guardian. Εκεί φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα ότι είναι ε, ε, μέλη σε μια εταιρεία χαρτοφυλακίου. Μόνο στην Ουγγαρία βρίσκεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμεί έχουμε μια κυβέρνηση συντηρητική, η οποία προασπίζεται χριστιανικέ αξίε και θέλει να παίζει σημαντικό ρόλο και στην εθνική πολιτική. Είπατε ότι το Ινστιτούτο τη Φλωρεντία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την συγκριτική μελέτη. Όμω το Ουγγρικό Media Institute έχει κάνει μια σχετική ανάλυση και ε, ελέγχθη ε, αυτό το κέσμα, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, έχω ακόμη ε, μισό λεπτό. Είναι σημαντικό να πω ότι βελτιώθηκε η κατάσταση τώρα σύμφωνα με το Ουγγρικό αυτό Ινστιτούτο και καταλήγουν τα μίδια να φτάνουν και 3 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα ε, ε, ακούν και μέσα τα οποία είναι επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Ενώ υπάρχουν άλλα όπως ε, στην τηλεόραση της RTL, η οποία έχει πρόσβαση σε πολλοί κόσμο. Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης μάλιστα στέκονται επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν είναι λοιπόν διόλου δίκαιο να πει κανείς ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο τα μέσα ενημέρωση της αντιπολίτευσης ή τα αντιπολιτευόμενα στην ε, Ουγγαρία. Κάποιοι περιορισμοί υπάρχουν. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εσείς, κυρία Αμπαμόντε, τώρα θέλετε να απαντήσετε. Μάλιστα, πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα, κυρία Ροσκόρ, για τη, Βοσκόρ, μάλλον, για την... Μπορείτε να μου στείλετε, αν θέλετε, τα πορίσματα της έρευνας του Ουγγρικού Ινστιτούτου. Ο Media Monitor εκδίδεται κάθε χρόνο. Αν θέλετε μπορώ να σα διαβιβάσω τα ευρήματά του. Βεβαίω οι κίνδυνοι δεν διαπιστώνονται μόνο στην Ουγγαρία. Βλέπουν τέτοιου και στην Ιταλία, στην Γερμανία, σε όλε τι χώρε μέλη. Στην πραγματικότητα. Αυτό που ζητήσαμε εν προκειμένου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω τη εξελίξεω αυτή και τη συγκεκριμένη αυτή ε, δημιουργία αυτού του ε, ομίλου, είναι μια ακόμη μελέτη η οποία θα συμπληρώσει τα πορίσματα της έρευνας του 2017. Και πάλι ε, τρέχοντος του έτους θα εκδοθεί και νέος Media Monitor που θα καλύπτει όλες τις χώρες μέλη. Αν επιθυμείτε μπορείτε να μου διαβιβάσετε τα πορίσματα της έρευνας του Ουγγρικού Ινστιτούτου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε τα μίντια είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Το ξέρουμε. Και γι' αυτό κάθε κυβέρνηση έχει και κάποια τάση να επηρεάζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ως πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες, τα γνωρίζουμε αυτά. Τα κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου αλλά και οι Εθνικές Βουλές, οφείλουν να σέβονται και να προασπίζονται την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά γιατί δεν αναφέρεστε και στην τσεχική δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργό. υπακούει στα ισχυρότερα μέσα της ε, τσεχικής δημοκρατίας. Είχαμε συζήτηση σχετικά στην ε, ε, Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και ακούσαμε εκεί και δημοσιογράφους από τα τσεχικά μέσα στενοχωριούμε πολύ που δεν έχουμε κανέναν δημοσιογράφο από την Ουγγαρία για να καταθέσει σχετικά με την κατάσταση των ε, μέσων. Και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόζουμε ίδια μέτρα και σταθμά για όλους. Ευχαριστώ. Σήμερα στη μερίσια διάταξή μας έχουμε την κατάσταση στην Ουγγαρία και νομίζω δικαίως, διότι υπάρχουν εκεί κάποιες πράγματι ανισχυτικές εξελίξεις. Γνωρίζουμε επίση, και ο κ. Αμπαμόντε το ε, τόνισε κατ' επανάληψη, ότι υπάρχουν και σε άλλε χώρε μέλη κάποιε ανισχυτικέ εξελίξει. Γι' αυτό και είναι σημαντικό, ακόμη σημαντικότερο για μα, η Επιτροπή μα να εγκύψει σε θέματα πολυφωνία των μέσων στι διάφορε χώρε μέλη. Και βεβαίω οφείλουμε να μετρούμε πάντοτε με ίσα μέτρα και σταθμά. Και μια φράση ακόμη για την RTL. Το γεγονό ότι η RTL στην Ουγγαρία. Είναι ένας από τους λίγους σταθμούς που επιτρέπεται ακόμη να ε, λειτουργούν και με επικριτικό τρόπο, το οφείλουμε στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε ε, ανάγκασε την Ουγγαρία να αλλάξει το νόμο περί ε, φορολογίας, διότι αλλιώς η RTL δεν θα μπορούσε πλέον να εκπέμπει από την Ουγγαρία, διότι δεν θα άντεχε οικονομικά. Τόσο απλό είναι. Δείχνει αυτό μάλιστα πόσο αναγκαίο είναι να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και εκεί και όχι μόνο στην Ουγγαρία, αλλά οπουδήποτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, διότι η πολυφωνία των μέσων, όπως γνωρίζουμε όλες και όλοι, είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας. Και πρέπει όλες και όλοι να φροντίσουμε ώστε να είναι εγγυημένη η ελευθερία αυτή και να επιτρέπει την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος μέσα σε πλήρη ελευθερία όπως ε, οφείλει που είναι στο κάτω-κάτω τύπος και τέταρτη εξουσία. Μήπως μπορεί, ε, λέει η κυρία να φτιάξει μια επισκόπηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι διάφορε μελέτε που γίνονται από το Media Center, ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα για ποιες χώρες μιλούμε, πώς, ε, ε, πώς εξελίσσεται η κατάσταση και μάλιστα όχι μόνο μέσα σε ένα έτος αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Να δούμε ποιες τάσεις διαμορφώνονται. Ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διαβάσει κάτι τέτοιο. Η κυρία Σαρτζεντίνη, ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνει δυνατότητα να κάνω ερωτήσει. και ευχαριστώ ιδιαίτερα που το θέσατε στην ημερήσια διάταξη. Πολλά ακούω. Θέλω να πω στους συναδέλφου ότι σύντομα θα μπορέσετε να ψηφίσετε στην Ολομέλεια για να ψήφισμα για την κατάσταση στη Σλοβακία και τη Μάλτα λόγω του θανάτου αυτών των δύο δημοσιογράφων που έκαναν έρευνες και ελπίζω να μας στηρίξετε. Και από πλευράς ε, και άλλων συναδέλφων θέλω να μάθω Τι δυνατότητε υπάρχουν να δουν τα θέματα ανταγωνισμού στην Επιτροπή. Λέτε πως ε, αν δεν μπορείτε από πλευράς ανταγωνισμού, ίσως μπορείτε να δείτε το θέμα των ε, δημοσίων βοηθειών. Γιατί όποια μέσα λαμβάνουν ε, κρατικές βοήθειες έχουν κάποιες υποχρεώσεις για πολυφωνία και ανεξαρτησία. Και κάτι ακόμη. Οι ιδιοκτήτες των μέσων ε, επεκτείνουν, της Ουγγαρίας επεκτείνουν και αλλού τις δραστηριότητές τους και στη Σλοβενία και στην ε, Μακεδονία. Τα εξετάζετε και αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Αμπραμόντε, Βεβαίω να σας στείλω τα στοιχεία ε, αυτό του Media Monitor που καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και αν έχουμε και στοιχεία από την Επιτροπή της Βενετίας και αυτά να σας τα στείλω, βεβαίως. Τι δυνατότητες έχουμε τώρα. Έχετε δίκιο. Ο κανονισμός για τις συγχωνεύσεις δεν λειτουργούν. Δεν ε, λειτουργεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί δηλαδή. Και δεν αναφέρεται υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εξαιρεθεί μία συγχώνευση από τα μέτρα κατά των μονοπωλίων αλλά οι κανόνες για τις κρατικές βοήθειες, ε, για, τις, ε, για τα καρτέλ, για το πώς μπορεί να στρεβλωθεί η αγορά λόγω κρατικών επιδοτήσεων, όλα αυτά ισχύουν. Θα σας ενημερώσω αφού μιλήσω με τους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ ανταγωνισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή τώρα. Δεν νομίζω να μιλούμε για τελευταία φορά για το θέμα αυτό και ιδίω για την Ουγγαρία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Αναμένουμε βεβαίω με ενδιαφέρον τι εργασίε του Ινστιτούτου τη Φλωρεντία και ασφαλώ θα παρακολουθούμε όλε τι εξελίξει, ιδίω όπω είπα στην Ουγγαρία και από ό,τι κατάλαβα από τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσεί θα πράξετε το ίδιο βεβαίως όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά όπου γύρονται κίνδυνοι κατά της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ε, σε μια πρώτη φάση μας ε, ενημερώσατε για τις εξελίξεις και θα είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες εάν μας ενημερώνετε τακτικά και να μας ε, διαβιβάσετε και τα ε, πορίσματα της έρευνας του Ινστιτούτου της Φλωρινδίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα παρακαλέσω όλες και όλοι όσοι δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δεν